Uh, uh, Ξεκινήσουμε. Έγκριση τη ημερήσιας διαταξής, αντιρρήσεις, ε, σχόλια όχι. Ωραία. Εγκρίνεται το σχέδιο ημερήσιας διάταξης χωρίς καμία αλλαγή. Σήμερα έχουμε όλες τις γλώσσες εκτός από την Κροατική. Θα ήθελα ακόμη μια φορά να σας υπενθυμίσω πως στις 3 και 4 ε, Φεβρουαρίου έχουμε την ε, κοινοβουλευτική εβδομάδα και μια εκδήλωση θα έχουμε την συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής στις 3 ε, Φεβρουαρίου 11 και 4 με μια η ώρα και η αίθουσα θα είναι πι 1α02. Και ελπίζω να έρθετε όλοι. Καλώς ήρθατε. Περνάμε μετά στο σημείο 3. Λάβαμε μία απόφαση. Οι συντονιστές πριν από τα Χριστούγεννα να προσκαλέσουμε να στηρίξουμε την ε, πρωτοβουλία του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας να μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα της ερευνητικής εργασίας ε, σχετικά με τον αντίκτυπο που θα έχει στην απασχόληση το επενδυτικό σχέδιο που παρουσίασε ο πρόεδρος της Επιτροπής. Ορίστε λοιπόν, έφτασε η στιγμή και δίνω τον λόγο στον κύριο Τόρες ο οποίος θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα κυρίες και κύριοι βουλευτές. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που δίνετε στον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας να παρουσιάσει την έρευνα αυτή για μια εκτίμηση του πιθανού αντικτύπου στην απασχόληση του επενδυτικού σχεδίου που ανακοινώθηκε. Ξεκινάμε βεβαίως με μια ανάλυση της κατάστασης στην Ευρώπη, την οποία γνωρίζετε. Έχουμε μια χαμηλή οικονομική ανάπτυξη και οι, προθε... προβλέψεις αναθεωρούνται προς τα κάτω, όπως βλέπετε τα βέλη προς τα κάτω, κόκκινα, οπότε οι προβλέψεις για οικονομική ανάπτυξη του 2015 αναθεωρούνται προς τα κάτω. 1,5% είναι η πρόβλεψη για φέτος σε σχέση με το πάνω από 3% στις ΙΠΑ και λιγότερο από ό,τι στις προηγούμενες προβλέψεις. Η κατάσταση επίσης χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλή ανεργία και βεβαίως ε, η ενεργεία στο 10% είναι πολύ ψηλότερη από ό,τι ήταν στην αρχή της κρίσης και υπάρχει και απόκληση μεταξύ ΕΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, κάτι το οποίο επίσης είναι γνωστό και αυτό δείχνει πως υπάρχει χαλάρωση της ε, χρήσης των δυνατοτήτων που υπάρχουν στην Ευρώπη. 23 εκατομμύρια άνθρωποι είναι άνεργοι και βεβαίω το βασικότερο εδώ πέρα είναι η μακροχρόνια ανεργία. 12 εκατομμύρια άνθρωποι είναι ανεργοί για πάνω από ένα έτος, δηλαδή μιλάμε για 40-50% και περισσότερους σε κάποιες χώρες. Κάτι το οποίο είναι σημαντικό, γιατί όσο περισσότερο μένει ο κόσμος άνεργος, τόσο πιο δύσκολο είναι μετά να ξαναμπεί στην αγορά εργασίας. Ένα σημαντικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η κατάσταση αυτή δείχνει πως υπάρχει έλλειμμα ζήτηση συνολικής ε, στην Ευρώπη, όχι μόνο λόγω των αριθμών της ανεργίας, αλλά γιατί η Ευρώπη και ειδικά η Ευρωζώνη έχει πλεόνασμα στους ε, εξωτερικούς ε, λογαριασμούς, κάτι το οποίο σημαίνει πως αποταμιεύει πολύ περισσότερα από όσα ξοδεύει η Ευρώπη. Ακριβώς λοιπόν είναι εδώ πέρα το έλλειμμα της ζήτησης στην Ευρώπη. Κάτι άλλο το οποίο είναι σημαντικό είναι πως πέρα από το έλλειμμα ζήτησης είναι πως τα παραδοσιακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για αυτή την κατάσταση δεν είναι τόσο χρήσιμα εδώ πέρα. Υπάρχει η λεγόμενη παγίδα ρευστότητα, δηλαδή τα επιτόκια είναι πάρα πολύ χαμηλά και πλέον δεν είναι αποτελεσματικά στο να κινητοποιήσουν επενδύσεις ή κατανάλωση λόγω της παγίδας ρευστότητας και είναι πάρα πολύ δύσκολο με αυτά τα συμβατικά μέσα μακροοικονομικής πολιτικής να επανεκκινήσει η οικονομία. Ο κίνδυνος βεβαίως είναι εδώ πέρα ο κίνδυνος αποπληθωρισμού. Έχοντας αυτά κατά νου, η προσέγγιση που έχουμε στην Ευρώπη ήταν να προωθήσουμε τις επενδύσεις μέσω του επενδυτικού σχεδίου και σε γενικές γραμμές βεβαίως αυτό θα ήταν χρήσιμο γιατί θα συμπλήρωνε την προσέγγιση που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξαιρετικά και συμβατικά νομισματικά μέτρα. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά είναι έμεσα μέτρα για να προωθηθεί η ζήτηση, γιατί η ζήτηση σχετίζεται με τις δαπάνες και ειδικά τις επενδυτικές δαπάνες. Οπότε το επενδυτικό σχέδιο είναι ένας άμεσος τρόπος να εκκινήσει η οικονομία με το να δοθούν κάποια κίνητρα για τις επενδύσεις. Και βλέπουμε εδώ πέρα στη ΣΥΠΑ πως ε, το χάσμα στην ανεργία εξηγείται σε σχέση με τις επενδύσεις. Οι επενδύσεις της ΕΠΑ έχουν ουσιαστικά φτάσει στα επίπεδα προ-κρίσης. Ένα 20% του ΑΕΠ επενδύεται. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι πολύ πιο χαμηλά από το επίπεδο προ-κρίσης. 17% του ΑΕΠ, ε, δηλαδή 3% κάτω από το επίπεδο προ-κρίσης και η τάση αυτή είναι προφανή στις χώρες με υψηλή ανεργία, στην ε, Νότια Ευρώπη, αλλά και με χαμηλή ανεργία, όπως στη Γερμανία. Οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι πιο χαμηλές από ό,τι ε, στο παρελθόν. Η ιδέα αυτή λοιπόν της ε, στήριξης απασχόλησης μέσω των επενδύσεων είναι σημαντική γιατί αντιμετωπίζουμε ακριβώς ε, την ρίζα του προβλήματος, ε, την έλλειψη ζήτηση, αλλά με επενδύσεις οι οποίες θα δώσουν δυνατότητα στην ευρωπαϊκή οικονομία να αναπτυχθεί και να δημιουργήσει δουλειές στο μέλλον. Ένα πάρα πολύ χρήσιμο μέσο. Στη μελέτη επίσης ε, βλέπουμε πως ε, το επενδυτικό σχέδιο θα μπορούσε να έχει είτε αμελητές ε, είτε σοβαρές επιπτώσεις ανάλογα με το πώς θα σχεδιαστεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες λοιπόν που έχουμε, το επενδυτικό σχέδιο έχει δύο στοιχεία. Το ένα είναι 63 δισεκατομμύρια ευρώ νέων, εάν θέλετε, επενδύσεων, δηλαδή 0,4% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και ένα άλλο στοιχείο, πολύ μεγαλύτερο, οι ιδιωτικές επενδύσεις, 252 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα σύνολο δηλαδή 315 δισεκατομμυρίων ευρώ, γύρω στο 2% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Αυτά και τα δύο μαζί λοιπόν είναι σοβαρά. Και αυτό βεβαίως πρέπει να το συγκρίνουμε με το επενδυτικό σχέδιο των ΙΠΑ, ανέφερα πριν τα νούμερα, που ήταν γύρω στο 5% του ΑΕΠ, ε, το διπλό δηλαδή, αλλά βεβαίως ε, κάπως πιο ε, μακροχρόνιο, αλλά συγκρίσιμα ποσά, αν όντως επενδυθούν πάνω από 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Οπότε η επένδυση αυτή για να ε, γίνει πραγματικά, να μεταφραστεί σε πραγματικές επενδύσεις στην οικονομία υπάρχουν δύο όροι. Ο ένας όρος είναι να συμβούν οι επιπρόσθετες επενδύσεις, οπότε η επιλογή των ιδιωτικών επενδυτικών έργων για το σχέδιο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική. Εάν οι επενδύσεις αυτές δεν επιλεγούν σωστά, αυτό το οποίο μπορεί να συμβεί είναι πως ε, θα υπάρχουν κάποιες επενδύσεις οι οποίες θα γινόταν ακόμα και απουσία του σχεδίου. Δηλαδή ε, θα έχει ελάχιστη, ελάχιστο επιπρόσθετο αποτέλεσμα. Και βλέπουμε ότι σύμφωνα με, τις, ε, με τους υπολογισμούς μας ε, σε αυτή την περίπτωση θα δημιουργηθούν μόνο 400.000 νέες θέσεις εργασίας μέχρι το 2018 που είναι ο χρονικός ορίζοντας του σχεδίου. Αντιθέτως, Εάν εκτελεστεί σωστά το σχέδιο, δηλαδή με μια προσεκτική επιλογή των έργων, υπολογίζουμε πως ο αντίκτυπος στην απασχόληση θα είναι 2,1 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας μέχρι το 2018, που θα επιτρέψει μία μείωση του ποσοστού ανεργίας κατά 1%. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι νομίζω θετικά νέα για την Ευρώπη. Η προσεκτική άρα επιλογή των επενδύσεων έχει κρίσιμη σημασία και πάλι εδώ πέρα η σημασία των νέων, καθαρών νέων επενδύσεων για να έχουμε καθαρά αποτελέσματα. Ε, διασυνδέσεις χωρών, ε, έργα, υποδομών, πράσινες επενδύσεις οι οποίες δεν θα γινόταν από ιδιώτες μόνο γιατί υπάρχει μια σημαντική διάσταση κλίμακας. Το άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό πέρα από την δικτύωση βεβαίως είναι η εμπλοκή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτές είναι βεβαίως έντασης εργασίας και μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις, ειδικά στις χώρες υψηλής ανεργίας, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν ε, προβλήματα λόγω της έλλειψης πίστοσης. Οπότε ε, μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες έχουν την δυνατότητα να αναπτυχθούν, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, αλλά δεν μπορούν λόγω της κατάστασης του πιστοτικού συστήματος σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Οπότε πρόκειται για, απασχόληση, για μεγιστοποίηση της επίδρασης στην απασχόληση και βεβαίως εκεί πέρα παίζουν σημαντικό ρόλο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και υπάρχουν ήδη κάποια παραδείγματα για το τι μπορεί να γίνει. Ξέρουμε παραδείγματο χάρη πως σε χώρες όπως η Δανία ή η Γερμανία υπάρχει ένα σύστημα εγγυήσεων πιστώσεων το οποίο επιτρέπει την εμπλοκή μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γνωρίζουμε επίσης πως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει κάποια εμπειρία στην εμπλοκή μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε επενδυτικά έργα. Αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής πάρα πολύ και πράγματι αυτά τα οποία έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέχρι στιγμής ε, εστιάζονται περισσότερο σε επενδύσεις γενικώ, γι' αυτό κάποιες από τις χώρες με υψηλή ανεργία έλαβαν λιγότερα δάνεια από την Ευρωπαϊκή ε, τράπεζα Επενδύσεων σε σχέση με χώρες με χαμηλή ανεργία. Παραδείγματο χάρη στην ε, Πορτογαλία βλέπουμε πως ε, επειδή ακριβώς έχει, έχουν κινητοποιήσει πλήρως τα κονδύλια Και βεβαίως υπάρχει αυτό το θέμα της δικτύωσης με άλλα έργα και βεβαίως το τι γίνεται με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επιπροσθέτως υπάρχει το ευρύτερο πλαίσιο και θεωρούμε ιδιαίτερα πως ε, οι πολιτικές ε, ενεργητικής ε, παρέμβαση στην αγορά εργασίας και άλλες θα μεγιστοποιήσουν τα ωφέλη του επενδυτικού σχεδίου και υπάρχουν εκτιμήσεις για 2,1 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας ε, εάν εφαρμοστούν αυτά και βεβαίως ε, κάτι άλλο σημαντικό είναι η αποκατάσταση της σχέσης μεταξύ της ε, σχέσης του εισοδήματος εργασίας και αύξησης της παραγωγικότητας. Οπότε η αποκατάσταση αυτής της σχέσης βεβαίως θα χρειαστεί περισσότερο καιρό, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική για να αναπτυχθεί ξανά η Ευρώπη. Και έτσι θα έχουμε άλλο ένα σημαντικό στοιχείο. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω πως μίλησα πολύ για το θέμα αυτό και για τις εκτιμήσεις και σας ευχαριστώ και πάλι για την ευκαιρία που μου δώσατε. Η ευκαιρία αυτή είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο αλλά και στην ιστοσελίδα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank Σας ευχαριστούμε και εμείς κύριε Τόρες. Είστε διευθυντής του Τμήματος Ερευνών στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εργασίας, Παγκόσμιο Οργανισμό Εργασίας. Έχω ορισμένου εγγεγραμμένους συναδέλφους. Θα αρχίσουμε τον Χάιντς Πέκε, ο οποίος ε, αντικαθέτων τον κύριο Κάς. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Τόρες. Μας δώσατε πληροφορίες για το λεγόμενο πακέτο Juncker. Μας φαίνονται σημαντικές. Επιθυμώ να τονίσω ιδιαίτερα ότι η βάση της επιτυχίας του πακέτου πρέπει τουλάχιστον αν κατάλαβα καλά αυτά που είπατε, να οριστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνει η καλύτερη δυνατή επιλογή των επενδυτικών έργων, έτσι ώστε να επιτευθεί και το maximum effect, αν θέλετε, στην απασχόληση. Ε, συγκεκριμένη ερώτηση λοιπόν. Πόσο αποτελεσματική θεωρείτε τον τρόπο, θεωρείτε, πόσο αποτελεσματικό μάλλον θεωρείτε τον τρόπο επιλογής των επενδυτικών έργων που από ό,τι βλέπω γίνεται καταρχήν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δεύτερο, δεύτερο ερώτημα, ποια θα ήταν κατά τη γνώμη σας τα ορθά κριτήρια για την βέλτιστη δυνατή επιλογή ενός επενδυτικού έργου με την έννοια της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα κριτήρια, υπάρχουν και άλλοι στόχοι ενδεχομένως για παράδειγμα, επιστροφή από επενδύσεις, return on investment, μπορεί να είναι πολύ σημαντικός στόχος αυτός. Βέβαια και εμένα με ενδιαφέρουν κυρίως οι στοχεύσεις εκείνες που θα επιτρέψουν τη δημιουργία του μέγιστου δυνατού αριθμού θέσεων απασχόλησης. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιούτα Στάινρουκ. Ευχαριστώ κύριε Τόρες με τη σειρά μου. Ευχαριστίες και στην οργάνωσή σας για την σημαντική αυτή μελέτη που ενδιαφέρει και εμάς εδώ τους ευρωβουλευτές και που δείχνει για άλλη μια φορά πόσο σημαντικό είναι και εμείς μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λαμβάνουμε υπόψη την πτυχή της απασχόλησης διότι σφάλματα που γίνονται ενδεχόμενα στο σχεδιασμό των επενδύσεων μπορούν να οδηγήσουν και σε λάθος αποτελέσματα. Διότι 1,8 εκατομμύρια βιώσιμες θέσεις απασχόλησης θα πρέπει να είναι και δικός μας στόχος για να ωφεληθούν οι πολίτες στην Ευρώπη. Και πρέπει να φροντίσουμε όλες και όλοι μαζί οι επενδύσεις αυτές να μην εκτοπίσουν τις ιδιωτικές επενδύσεις, διότι τότε χάνεται αυτό το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα και εσείς είπατε ότι μπορούν να υπάρξουν και αντίθετα αποτελέσματα εάν το πακέτο αυτό επενδύσεων γίνει και αντικείμενο λανθασμένων χειρισμών. αλλά και να γίνουν στοχευμένες επενδύσεις στις χώρες εκείνες μέλη που σημειώνονται τα μεγαλύτερα προβλήματα και όπου η ανεργία των νέων είναι μεγαλύτερη, όπου είναι ανάγκη να αντιμετωπιστεί η μακροχρόνια ενεργεία. Αυτά λοιπόν να είναι δεσμευτικοί στόχοι του πακέτου. Τώρα, ερώτηση, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ώστε στις χώρες όπου σημειώνονται τα μεγαλύτερα προβλήματα, που χρειάζονται και τη μεγαλύτερη υποστήριξη, εκεί να γίνουν οι επενδύσεις αυτές. Στη μελέτη σας έχετε καταλήξει συμπεράσματα για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Ταμείο Επενδύσεων έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί και μάλιστα σε βάθος χρόνου η ανεργία των νέων. Ευχαριστώ. Γεια σου Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για αυτή την παρουσίαση. Είναι, ήταν διεξοδική. Ιδίω η παρουσίαση στοιχείων ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, όμως έχω κάποιες αμφιβολίες για τα κονδύλια και ίσως μπορείτε να με βοηθήσετε σε σχέση με τι απορίε που έχω. Το Ταμείο θα απευθύνεται από τη μια στι μικρομεσαίε επιχειρήσει και από την άλλη επενδύσει. συνήθω ήταν μεγάλη κλίμακα στη διαδικτύωση, στι μεταφορέ Το Ταμείο σκοπό έχει να κινήσει ε, ενεργητικό, στοιχεία του ενεργητικού που αυτή τη στιγμή έχουν παγώσει προ τι επενδύσει. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει θα μπορούν να τα υλοποιήσουν αυτά τα μεγάλα σχέδια και προγράμματα. Αυτά τα παγωμένα στοιχεία του ενεργετικού που δεν χρησιμοποιούνται για τι επενδύσει αυτή τη στιγμή θα αξιοποιηθούν από τι μικρομεσαίε. Αυτή είναι η πρώτη μου απορία. Και η δεύτερη είναι πώ το... θα διαχειριστούμε το Ταμείο. Συζητούμε ότι πρέπει να επιλέξουμε τα καλύτερα προγράμματα. Όμω, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διευθυντική αυτή Επιτροπή που θα δημιουργηθεί που θα ιδρυθεί και θα διαχειρίζεται το Στατηγικό Ταμείο Επενδύσεων μπορεί να έχει και πολιτικές διαστάσεις, πολιτικό χαρακτήρα. Πώς θα αποφύγουμε να γίνει ένας πολιτικός φορέας στο Ταμείο αυτό. Επίσης λέμε ότι στην Διευθύνουσα αυτή η Επιτροπή θα συμμετέχουν ε, πρόσωπα που εκπροσωπούν αυτούς που συνεισφέρουν τα περισσότερα στο Ταμείο. Αυτό το έχετε εξετάσει. Πώς θα αποφύγετε να λάβει πολιτικές διαστάσεις στο Ταμείο. Ευχαριστώ κύριο Στόμασμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για τη μελέτη. Χρήσιμη μου φαίνεται. Είπατε ότι μάλλον εξοικονόμηση γίνεται σε πολλούς τομείς παρά επενδύσεις. Σωστό είναι αυτό. Πολλοί όμως διερωτώνται, αξίζει να επενδύσω άμα δεν ξέρω τι μέλλον θα έχει επένδυση. Αυτό ισχύει και για επιχειρήσεις που προσπαθούν και πέραν από τα όρια των χωρών τους, κυρίως οι μικρές και μισές επιχειρήσεις μιλώ εδώ, όπου τους καταστήσαμε δυνατό με την Enterprise για να μπορούν να συνεργαστούν. Αλλά όλα αυτά είναι, πώς να το πω, τρυφερά βλαστάρια. Δεν είναι βέβαιο ότι θα επιβιώσουν. Ρώτησε κάποιος άλλος πριν τι πιθανότητες έχουν να πετύχουν οι επιχειρήσεις αυτές. Είναι σημαντικό αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ότι δηλαδή ε, αυτό το Διευθυντικό Συμβούλιο το οποίο ε, δεν θα είναι πολιτικό, θα, είναι, θα αποτελείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που θα μπορούν να αξιολογούν τα, τις επενδύσεις. Τι γίνεται όμως, ποια εγγύηση υπάρχει όταν θα κάνουν την επιλογή θα μπορούμε να γνωρίζουμε ότι αυτό το επενδυτικό σχέδιο τελικά θα υιοθετηθεί ή θα αναλαμβάνουν πλέον οι χώρες μέλη, θα εξετάζουν την πρόταση των εμπειρογνωμόνων και θα αρχίζει μετά το γνωστό παζάρι. Δώσε με αυτό για να σου δώσω εκείνο. Το χειρότερο θα είναι αυτό, διότι θα καταλήξουμε τότε σε επενδυτικά σχέδια που δεν θα έχουν απολύτω καμία ουσία, καμία προστιθέμενη αξία και δεν θα ληφθεί καθόλου υπόψη εκεί η διάσταση τη απασχόληση. Δηλαδή κάποια παλιά σχέδια τα οποία κάπως θα ωρεοποιηθούν με ευρωπαϊκά χρήματα. Τώρα, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να προσελκύσουμε ιδιωτικά κεφάλαια. Πού να επενδύσουν όμως αυτά. Θέλουμε κάτι να μπορεί να προκύψει από την επένδυση αυτή. Όπου σημειώνονται δυσκολίες στην απασχόληση να υπάρξουν επιτυχίε, δηλαδή συγκεκριμένε επιτυχίε Με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχουμε πετύχει ορισμένα πράγματα. Αλλά χρειάζεται, υπάρχουν δηλαδή τα κριτήρια αξιολόγηση Έχω όμω τι αμφιβολίε μου εάν εν τέλει θα οδηγηθούμε σε κάποιο αποτέλεσμα που να μπορεί να πει κανεί ότι το αποτέλεσμα αυτό είναι αρκετά αντικειμενικό και δεν θα μπει μέσα σε ένα πολιτικό καυγά τελικά. Ευχαριστούμε Μαρία Ζωάου Ροντρίγκεφ. Κύριε Τόρες, ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Πολύ επίκαιρη και πολύ ενδιαφέρουσα για να ε, εμπλουτίσει την ευρωπαϊκή συζήτηση. Βρίσκω την εζωτική σημασία στη συζήτηση για μας στο Κοινοβούλιο και αυτή την Επιτροπή. Και είναι πολύ ωραίες οι ιδέες που μας δώσατε για τα κριτήρια επιλογής των προγραμμάτων. Επιτρέψτε μου να τονίσω τρία από τα κριτήρια. Πρώτον, οι στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις επενδύσεις ώστε να υπάρξει μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης. Δηλαδή να δώσουμε προτεραιότητα σε προγράμματα που συνάδουν με την μετάβαση των ενεργειακών μας προτεραιοτήτων, της των ψηφιακών προτεραιοτήτων μαζί με κοινωνική ένταξη και των κοινωνικών επενδύσεων την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, του ανθρώπου. Εδώ μπορούμε να, να δημιουργήσουμε πολλέ θέσει απασχόληση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τι κοινωνικέ υπηρεσίε ή τι υγειονομικέ. Δεύτερο κριτήριο και το αναφέρατε είναι η διασύνδεση της Ευρώπης το Connecting Europe. Θα πρέπει να καλύψουμε τις ελλείψεις που έχουμε στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Υπάρχει όμως και ένα τρίτο κριτήριο να μειώσουμε τις μακροοικονομικές ανισότητες. Εκεί πρέπει να χρησιμοποιήσουμε επενδύσεις ώστε να καλύψουμε αυτή τη ε, διαφορά στις μακροοικονομικές ε, συνθήκες των κρατών μελών διότι ακριβώς είναι πολύ διαφορετική όρη επενδύσεων των κρατών μελών και αυτό είναι ένα ζήτημα κεντρικής σημασίας για την Ευρώπη σε αυτή τη φάση. Νομίζω λοιπόν ότι οι επενδύσεις που θα σχεδιαστούν πρέπει αυτό να το έχουν ε, λάβει υπόψη στο σχεδιασμό. Ε, ξέρετε ότι στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων έχουμε μια πολύ έντονη συζήτηση για αυτό, διότι ως τώρα ο κανονισμός που μας ε, προσφέρεται δεν επιτρέπει ίσους όρους αξιοποίησης του Στατηγικού Ταμείου από τα κράτη-μέλη οι χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση δεν έχουν τους ίδιους όρους. Εάν αυτό το πρόβλημα δεν το ξεπεράσουμε, οι ανισότητες θα αυξηθούν και με την επενδυτική διαδικασία και όχι αντιστρόφως. Απλώς προς ενημέρωσή σας. Και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τον οργανισμό σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Τόρες. Σειρά σας possible. Πρώτα σας ευχαριστώ για τις αντιδράσεις που άκουσα για την μελέτη και την ανάλυση μας. Οι ερωτήσεις που κάνετε βέβαια είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Πρώτα, πώς να αναμειχθεί η Ευρωπαϊκή, και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Ρωτήσατε επίσης πολύ για τα κριτήρια επιλογής των επενδυτικών έργων. Βεβαίως αυτά είναι η καρδιά του θέματος, γιατί εάν τα κριτήρια δεν είναι καλά καθορισμένα, υπάρχει ο κίνδυνος πάλι οι επιπτώσεις, οι θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση να είναι πολύ περιορισμένες. Μπορεί βέβαια να μπουν και άλλα μη οικονομικά κριτήρια ή η πολιτική ανάμειξη και να μην ε, μεγιστοποιηθεί το αποτέλεσμα στην απασχόληση. Για να μεγιστοποιηθεί το αποτέλεσμα στην απασχόληση, πιστεύω είναι βέβαιο ότι οποιοδήποτε επενδυτικό έργο πρέπει να έχει μια εξωτερικότητα και αυτά πρέπει να είναι πρώτη επιλογή. Δηλαδή θα είναι επενδυτικά έργα τα οποία δεν θα είναι επενδυτικά έργα τα οποία θα γίνουν με απουσία του επενδυτικού σχεδίου. Για την ανάπτυξη δικτύων στην Ευρώπη, για την ψηφιακή οικονομία, καθιστάμεθα μάρτυρες μιας νέας τεχνολογικής επανάστασης που σύμφωνα με τον ILO θα έχει βαθύτατες επιπτώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο και εξαρτάται από το πώς οι διάφορες χώρες θα αρπάξουν τις ευκαιρίες που ανοίγονται. Τα σενάρια για το μέλλον σε ό,τι αφορά την απασχόληση και την παραγωγικότητα θα είναι αντίστοιχα με αυτή την ικανότητα των χωρών πάρα πολύ διαφορετικά και θα εξαρτηθεί και από την ικανότητα τη Ευρωπαϊκή οικονομίας να αδράξει αυτές τις νέες ευκαιρίε για τη δημιουργία απασχόλησης που θα είναι θετική για την απασχόληση, θετική για τις επιχειρήσεις και για τη μελλοντική ευημερία της Υπήρου. Αυτά λοιπόν είναι σημαντικά κριτήρια. Εφόσον εφαρμοστούν σωστά τα κριτήρια αυτά, θα βελτιώσουν το επενδυτικό κλίμα, θα βελτιώσουν την επένδυση και επίσης και την επιστροφή από την επένδυση. Άρα χρειάζεται ισχυρή εξωτερικότητα, δηλαδή πράσινη οικονομία, επίσης το η ιδέα συνδέοντας την Ευρώπη, συνολικά οι συνδέσεις στην Ευρώπη, γιατί από μόνο το ένα επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να το επιτύχει αυτό. Το δεύτερο κριτήριο, και θα πρέπει να είναι ξεχωριστό, γιατί δεν έχει τον ίδιο χαρακτήρα, θα πρέπει να είναι ότι θα πρέπει να απευθύνονται σε μικρές επιχειρήσεις. Μπορούν να μπουν οι μικρές επιχειρήσεις σε αυτά τα μεγάλα project, αλλά συνήθως δεν θα το πράξουν. Εδώ λοιπόν, με σχετικά χαμηλά κονδύλια, μπορεί να προωθηθεί αυτή η ιδέα των εγγυήσεων πιστώσεων, ιδίω αυτά μπορούν να εξυπηρετήσουν χώρε όπου βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτό δείχνει η εμπειρία πάντω. Και πάλι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να γίνει το θεσμικό εκείνο όργανο που έχει αντίστοιχα στη Γερμανία και στη Δανία για παράδειγμα, που προσφέρει εγγυήσει πιστώσεων σε μικρές επιχειρήσεις που μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις ή οι τράπεζες αναλόγως και αυτό δίνει όθηση σε νέες επενδύσεις και επομένως στη δημιουργία απασχόλησης που δεν θα γινόταν αν δεν υπήρχαν αυτές οι εγγύησεις. Αυτό λοιπόν είναι ξεχωριστό είδος επενδυτικών ευκαιριών. Το άλλο είναι, ε, με ρωτήσατε για την πολιτική ανάμειξη εδώ, επιτρέψτε μου να μην επεκταθώ πολύ γιατί δεν είναι η ειδικότητά μου, θα πω μονάχα ότι στην έκθεσή μας τονίζουμε την ανάγκη monitoring και αξιολόγησης, ακόμα και για καλά καθορισμένα επενδυτικά έργα που καμιά φορά ξεφεύγουν από τον δρόμο που τους έχετε βάλει. Πρέπει λοιπόν να γίνεται παρακολούθηση του επενδυτικού έργου από την αρχή και βεβαίω να γίνεται αξιολόγηση. Η αξιολόγηση πρέπει να είναι βεβαίως δημόσια πολιτική, ιδίω όμως και για κάθε πολιτική βεβαίω, κάθε δημόσια πολιτική χρειάζεται ε, αξιολόγηση, αλλά ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια. Και η ανάμειξη στο monitoring και στην αξιολόγηση, η ανάμειξη μιας διάστασης της απασχόλησης. Άρα να μην αξιολογείται μονάχα ε, η απόδοση της επένδυσης, το return, αλλά και η υλοποίηση της διάστασης της απασχόλησης. Βεβαίως, εάν επιλεχθεί αυτή η προοπτική, αυτή η ε, προσέγγιση μάλλον, που εσείς θα το αποφασίσετε αυτό, θα είναι σημαντικό να την υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τώρα, ποια θα είναι η χρήση, ποια θα είναι η χρησιμότητα για τους νέους. Βεβαίω η ανεργία των νέων είναι πάρα πολύ ψηλή σε ορισμένες χώρες και αυτό είναι μεγάλη ανησυχία. Εσείς ήδη έχετε αποφασίσει να θεσπίσετε την εγγύηση απασχόλησης των νέων που δοκιμάστηκε στο χρόνο, για παράδειγμα στις ε, βόρειες οικονομίες των βόρειων χωρών, δηλαδή σκανδιναβικών κλπ. Δοκιμάστηκε αυτή η εγγύηση των νέων ήδη από τη δεκαετία του 90. Θα έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα το πρόγραμμα αυτό, θα συμβαδίζει χέρι με χέρι δηλαδή με το επενδυτικό σχέδιο, θα πρέπει όμως να αναβαθμιστεί, διότι η χρηματοδότηση που έχει σχεδιαστεί από τις χώρες ως τώρα είναι περιορισμένη. Χρειαζόμαστε λοιπόν περίπου 21 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο στην Ευρώπη για να είναι αποτελεσματική η ε, εγγύηση απασχόληση των νέων. Να είναι καλά εξοπλισμένες με προσωπικό, καλά στελεχωμένες δηλαδή οι αρμόδιες υπηρεσίες και αυτό θα αποτελέσει τότε ένα πολύ χρήσιμο συμπλήρωμα στο επενδυτικό σχέδιο γιατί αυτές οι υπηρεσίες θα επιτρέψουν την επανένταξη στην αγορά εργασίας των νέων ανθρώπων ή και την πρώτη εργασία, για παράδειγμα σε χώρους όπως της ψηφιακής οικονομίας, της πράσινης οικονομίας ή και σε άλλους κλάδους, ή μάλιστα να τους βοηθήσει να δημιουργήσουν και δικές τους δουλειέ, δικέ του επιχειρήσεις. Νομίζω ότι με τα λόγια αυτά κάλυψα τα περισσότερα για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, επίσης τα αποτελέσματα δικτύων, networking effects και πάλι για τις μικρές και μέσες επιχειρήσεις είπε η κυρία Ροντρίγκες ότι θα πρέπει ίσως να προσθεθεί ένα τρίτο κριτήριο που αναφέρεται στις μακροοικονομικές ανισορροπίες αλλά με λήψη υπόψη του ρόλου των μικρών και μεσών επιχειρήσεων και των connection effects, ήδη αυτό θα επιτρέψει σε ορισμένες χώρες να αποφεληθούν περισσότερο. Ίσως να πρέπει να ληφθεί υπόψη και το πανευρωπαϊκό στοιχείο του επενδυτικού σχεδίου. Επιπρόσθετα δηλαδή των κρατικών επενδυτικών στοιχείων, ε, σχεδίων. Και να δοθεί βέβαια περισσότερη προσοχή σε χώρες και σε τομείς όπου σημειώνεται μεγαλύτερη ανεργία υπάρχει ένα στοιχείο 20% αλληλεγγύης μέσα σε αυτή τη νέα πολιτική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ίσως το ίδιο πνεύμα μπορεί να λειτουργήσει και για να ε, αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο αυτό θέμα. Ευχαριστώ. Να προχωρήσουμε τότε με τις ερωτήσεις. Ο κύριος Σούλτσε, ευχαριστώ κύριε Τόρες. Συμφωνώ με πολλά από τα όσα είπατε και με συναδέλφους που σχολίασαν. Ξανά στις μικρές και μεσές επιχειρήσεις, διότι εκεί εργάστηκα ούτως ή άλλως για μια δεκαετία πριν να εκλογώ ευρωβουλευτής. Με εκπλήσουν καμιά φορά οι συζητήσεις αυτές, διότι φαίνεται ορισμένοι να πιστεύουν ότι ρίχνουμε λεφτά στην αγορά, βοηθάμε τις μικρές και, και μεσές επιχειρήσεις και ξεκινάει ξανά ο σειρμός. Όποιος τα πιστεύει αυτά κάνει λάθος, λάθος μεγάλο επειδή μου δίνετε μονάχα 2-3 λεπτά ε, χρόνο αγόρευσης, να σας πω ότι όχι μόνο στη Γερμανία, από την οποία προέρχομαι, αλλά και σε όλες τις ε, χώρες μέλη, έχουμε τρεις διαφορετικές κατηγορίες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Κάποιες οι οποίες αποδίδουν και αυτές δαν, δανειοδοτούνται ευκολότατα. Έχουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ε, πρέπει να πει κανεί ότι δεν τα καταφέρνουν και τόσο καλά, αλλά αξίζει να υποστηριχτούν και αυτέ λοιπόν λαμβάνουν χρήματα, διότι υπάρχουν λεφτά στην αγορά. Και υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία, και νομίζω αυτέ είναι οι πρώτε οι οποίε θα ρηχτούν πάνω στα project αυτά που συζητούμε, που δεν βρίσκουν λεφτά στην αγορά. Γιατί όμω όχι, και πού βρίσκεται το πρόβλημα, εκεί λοιπόν έχω σημαντικότατε επιφυλάξει. Δηλαδή να πάμε να δώσουμε υγιέ χρήμα σε μικρέ και μεσές επιχειρήσει για να τι υποστηρίξουμε δηλαδή, που το προϊόν τους στην αγορά δεν ενδιαφέρει κανένα. Να τις κρατήσουμε δηλαδή στη ζωή για 3, 4, 5 χρόνια και μετά, μετά από μια πενταετία να δούμε ότι οι επιχειρήσεις αυτές διαλύονται, εξαφανίζονται και ότι πρέπει να τις υποστηρίξουμε αν θέλουμε να διατηρηθούν μονάχα με χρήματα των φορολογουμένων, με ενέσεις από χρήματα των φορολογουμένων. Ίσως λοιπόν με τα χρήματα αυτά να κάνουμε καλύτερα επενδύσεις σε εκπαίδευση στα μυαλά των ανθρώπων, γιατί τότε θα βελτιώσουμε και την θέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που τώρα δεν διασώζονται όσα λεφτά και να τους διαθέσετε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια χώρα όχι μόνο όπως η Γερμανία που σε αυτό το τομέα τα καταφέρνει, αλλά και για άλλες χώρες. Γι' αυτό ξαναλέω, επενδύσεις στα μυαλά των ανθρώπων. Εκεί χρειάζονται στην πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Κυρία Ζούμπερ. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Τόρες για την παρουσίασή του. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με το είδος απασχόλησης που μπορεί να δημιουργηθεί μέσω αυτού του προγράμματος. Και κάτι που πάει λίγο παραπέρα Το ποσοτικό θέμα επίσης, πόσες θέσεις μπορεί να δημιουργηθούν, διότι σήμερα μιλάμε πάρα πολύ με την ανάγκη, για την ανάγκη που ε, υπάρχει να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης, προφανώς, αλλά ξεχνάμε ότι ζούμε σε καιρούς που ούτως ή άλλως υπήρχε ανεργία. Αυτό που έλειπε ε, ο βασικά ήταν η ποιότητα στην εργασία, τα δικαιώματα τα εργατικά δικαιώματα. Εάν σκεφτούμε την εποχή της δουλείας, υπήρχε πολλή δουλειά, σίγουρα, αλλά χωρίς καθόλου δικαιώματα. Οπότε το ερώτημα που θέλω να θέσω έχει να κάνει με την προοπτική, με το τι διασφάλιση έχουμε από το πρόγραμμα, ότι θα δημιουργηθούν θέσει απασχόληση, αλλά και τι είδου θέσει, πώ θα έχουν κάποια βιωσιμότητα για το μέλλον. Δεν θα επιθυμούσαμε το πρόγραμμα αυτό να στηριχθεί από κάποιους μεγάλους ιδιωτικούς ομίλους, από ιδιωτικά ιδρύματα που ξέρουμε ότι μπορούν να κάνουν επενδύσεις, προφανώς, αλλά πέραν αυτού και μετά από αυτό, για τους εργαζομένους και τις ζωές τους, δεν μένει τίποτα στα χέρια. Ε, αυτή είναι η βασική μου ερώτηση, λοιπόν. Πώς μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι και να διαφυλάξουμε και να εγγυηθούμε ότι μέσα από το πρόγραμμα αυτό τα εργατικά δικαιώματα θα προστατευτούν και οι θέσει εργασία που θα δημιουργηθούν θα είναι αξιοπρεπεί και θα συνάδουν με τι κοινωνικέ μα προδιαγραφέ. Μόνικα Μάνερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστούμε τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας για την μελέτη αυτή. Είναι σημαντική συνεισφορά στο θέμα της δημιουργίας θέσεων εργασίας και να δούμε βεβαίως ε, τον αντίκτυπο που θα έχει το σχέδιο αυτό και να δούμε βεβαίως και την βιωσιμότητα των ε, θέσεων εργασίας αλλά βεβαίως και θα έπρεπε να είναι και κομμάτι του σχεδίου η αηφόρος ανάπτυξη. Επίσης βλέπουμε εδώ πέρα πως υπάρχει μια δυναμική την οποία πρέπει να εξαντλήσουμε και να δημιουργηθούν οι συνθήκες πλαίσιο για να εξαντληθεί όλη αυτή η δυναμικότητα. Τώρα, είπατε κι εσείς πως είναι ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση και χρειαζόμαστε πολλά περισσότερα μέτρα για να έχουμε πραγματικά μια πιο αηφόρο ε, οικονομία με περισσότερες δουλειές. Αλλά μιλήσατε για 400.000 ε, θέσεις εργασίας ως μίνιμουμ και το πιθανό maximum 2,1 εκατομμύρια υπό διάφορες προϋποθέσεις ε, όπως επένδυση στις περιοχές που έχουν μεγάλη ενεργεία, συνοδευτικά μέτρα, νέα έργα κτλ. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό το 300.000 που αναφέρατε ως minimum. Ε, είναι σίγουρα αυτά που μας λέτε έχετε λάβει ε, υπόψη διαφορετικά σενάρια και βεβαίως ε, το, για την ε, μόχλευση. Και επίσης πώς βλέπετε τους ε, κλάδους. Αλλά αναφέρατε βεβαίως πως η παραγωγικότητα είναι τελείως διαφορετική αν μιλάμε για ψηφιακή οικονομία ή για την πολεοδομία, πώς θα ζυγίζεται όλα αυτά. Αλλά όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, το θέμα δεν είναι μόνο να ε, δημιουργηθούν κάποιες θέσεις εργασίας, αλλά ποιες θέσεις εργασίας. Ε, μπορεί κάποιος να ζήσει από αυτές τις θέσεις εργασίας, είναι βιώσιμες ε, και βεβαίως θα πρέπει να δούμε ποιες ακριβώς είναι οι επιπτώσεις, να υπάρξει μια παρακολούθηση των επιπτώσεων. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε σαφείς στόχους, ειδικά στις κατευθυντήριες γραμμές, ε, στο Διοικητικό Συμβούλιο του έργου αυτού, να υπάρχει επίσης ε, η αρχή της εταιρική σχέσης με τις τοπικές αρχές, κοινωνικούς εταίρους, κοινωνία των πολιτών. Εκεί πέρα πρέπει να γίνουν πολλά σε πολιτικό επίπεδο ακόμα. Ευχαριστώ. Μπάλας. Πολύ γρήγορα διότι ουσιαστικά θα συνεχίσω αυτό που είπε η κυρία Ροντρίγκες προηγουμένως για τις διάφορες περιοχές της Ευρώπης και τις μακροοικονομικές ανισότητες, τις αποκλήσεις μεταξύ τους. Ε, σήμερα φαίνεται να είναι πιο έξυπνο να επενδύσουμε εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη αν και δεν θα πρέπει να τα κάνουμε τα πράγματα ε, να φαίνονται κομικά. Ακόμα και στην Γερμανία υπάρχει ανάγκη επενδύσεων, ακόμη και αν είναι μια μεγάλη χώρα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να βλέπουμε τα πράγματα ε, γραφικά. Υπάρχει ανάγκη επενδύσεων ακόμα και στις χώρες, στις μεγάλες χώρες της Ευρωζώνης. Όμως χρειάζεται και μια αλληλεγγύη ώστε να επιβιώσει το ενιαίο νόμισμα. Και αυτό είναι σημαντικό. Έχετε, και αυτό είναι το συγκεκριμένο με ερώτημα, στη μελέτη σας ε, στοιχεία για τις διαφορές ανάλογα με τις γεωγραφικές ζώνες και διαφορετικά σενάρια, διαφορετικές υποθέσεις. Συμφωνώ βεβαίως ως προς την ψηφιακή ατζέντα ή την ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Όμως τη γεωγραφική διάσταση την έχετε λάβει υπόψη και αν ναι, είναι το αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε κυρία Μπουλκεβιτσιούτα. Ε, ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστούμε για την μελέτη. Έχω μερικέ ερωτήσει. Πρώτα απ' όλα και πρωτίστως η απασχόληση και κοινωνικέ πολιτικέ. Έχουν άμεση σχέση με την οικονομία και τον αντίκτυπο των βιώνουν περισσότερο από όλους οι πολίτες. Όσοι δεν έχουν δουλειά, όσοι δεν έχουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Τα κίνητρα για τις επενδύσεις είναι επίσης πολύ σημαντικά. Πρέπει να μιλήσουμε και για κίνητρα λοιπόν, το είπατε κι εσείς. Θέλω να ρωτήσω ποιες, ποια συγκεκριμένα κίνητρα έχετε κατά νου και τι κίνητρα θα μπορούσαν να διασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις στα κράτη-μέλη θα είναι ε, βιώσιμες, διαρκείας και μακροχρόνιες και ότι θα υπάρξει πραγματικό κέρδος για τους πολίτες μας. Ίσως η κάθε χώρα να πρέπει να λάβει τις δικές της αποφάσεις ή μήπως πρέπει να υπάρξει κάποια απόφαση ευρωπαϊκή περί κινήτρων για τις επενδύσεις. Και μία ακόμη ερώτηση. Οι συνάδελφοι μίλησαν πολύ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι όντως πολύ σημαντικές για τις οικονομίες μας και την πολιτική απασχόληση, διότι δημιουργούν πολλές θέσεις. Όμως η ερώτηση, η βασική ερώτηση είναι γιατί οι μικρομεσαίες δεν λαμβάνουν πιστώσεις, δάνεια, ώστε να μπορέσουν επιτέλους να δημιουργήσουν αυτές τις θέσεις απασχόλησης. Γιατί, γιατί δεν έχουν πρόσβαση στις πιστώσεις. Ποιοι είναι οι λόγοι. Με το επενδυτικό πρόγραμμα θα λάβουν οι μικρομεσαίες πιστώσεις για να δημιουργήσουν θέσεις. Και μία ακόμη ερώτηση. 25 εκατομμύρια άνεργοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 12 εξ αυτών μεγάλης, μεγάλης διαρκείας ε, άνεργοι, επιμακρών άνεργοι. Εάν επενδύσουμε στην ενέργεια για την ψηφιακή οικονομία, σημαίνει αυτό ότι τα 25 εκατομμύρια άνεργοι θα καλύψουν αυτές τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν υπάρχουν αρκετά κίνητρα για να καλύψουν οι πολίτες αυτές τις θέσεις. Διότι έχουμε ανθρώπους που ξέρουν να δουλεύουν, που έχουν τις γνώσεις, που έχουν την απαραίτητη κατάρτιση. Οπότε το ερώτημα είναι εάν το επενδυτικό πρόγραμμα θα είναι πιο αποτελεσματικό εφόσον επικεντρωθεί στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων μας. Πολλοί είναι οι συνάδελφοι που σχολίασαν για τη μελέτη σας και είπαν πόσο επίκαιρη είναι. Δεν χρειάζεται να τα ξαναπώ κι εγώ, όσο και αν συμφωνώ. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια της δουλειάς του ILO, του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και έχω μια ερώτηση για ένα ζήτημα που μαζί με όλα τα άλλα έχει τεθεί Είχα εντατικές συνομιλίες με κάποιον από την ΕΤΕ που λέει ότι τώρα θα προσλάβουν περισσότερο προσωπικό, ότι χρειάζονται 500 άτομα για να δουν όλα αυτά τα νέα προγράμματα. Αλλά λένε, έχουμε και τους περιορισμούς μας για το τι, επιστροφή περιμένουμε από τις, ε, τι επιστροφές περιμένουμε από τις επενδύσεις. 18% περιμένουμε τη απόδοση. 18% ε, περιμένουμε. Αλλά εάν θέλει κανείς ε, τα προγράμματα με περιβαλλοντική διάσταση, ή με κοινωνική και δημιουργία θέσεων απασχόλησης, Λέει και η ΕΤΕ ότι για να επιλεγούν αυτά τα προγράμματα πρέπει και εμείς να καλύψουμε τις δικές μας ανάγκες απόδοσης. Δεν είναι λοιπόν ε, μια καθιερωμένη ε, διαδικασία για αυτούς. Ε, πρέπει να δουν πολλά νέα προγράμματα. Αλλά για τη δική τους τη μεθοδολογία <clears throat> δεν θα υπάρξουν προγράμματα αναγκαστικά που θα εμπλουτίζουν τις θέσεις εργασίας, που θα τις πολλαπλασιάζουν. Δεν θα είναι αυτό το κριτήριό τους. Ξέρετε εσείς ποια κριτήρια ακριβώς χρησιμοποιείτε σε σχέση με το στατηγικό ταμείο. Παλώμα Λόπες Περμέγιο. Ευχαριστούμε. Μιλήσατε για τη δημιουργία 1,8 ε, εκατομμυρίου θέσεων απασχόλησης. Ε, Όντω, ακούσαμε ότι θα υπάρχουν νέε επενδύσει, αλλά μέχρι τώρα δεν είναι και τόσο σοβαρέ με 23 δι. Σαν επιδότηση μοιάζει από την ΕΤΕ. Ε, όταν μιλάμε για τις ε, για τα προγράμματα, οι επενδύσει φαίνεται ότι θα γίνουν κυρίω σε χώρε που ήδη έχουν καλέ οικονομικέ επιδόσεις. Ήδη υπάρχουν επενδύσει. Άρα μακροχρόνια θα επικεντρωθείτε σε χώρες, θα επικεντρωθεί το πρόγραμμα σε χώρες που, που έχουν χαμηλή ενεργεία και υψηλή ανάπτυξη. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα δημιουργηθούν λιγότερες θέσεις απασχόλησης από ό,τι ευαγγελίζεστε, ε, λιγότερες από ό,τι ελπίζουμε. Οπότε να θυμίσω ότι η ΕΤΕ ήδη δυσκολεύεται να δαπανίσει όλα τα χρήματα που διαθέτει λόγω τεχνικών περιορισμών και πολιτικών αποφάσεων. Έχουν δοθεί πιστοτικές γραμμές σε προγράμματα που δεν έχουν πετύχει και πολύ λίγα δίνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τον ε, κλάδο αυτό. Ε, δύο ερωτήσεις λοιπόν. Τι είδους εγγύησεις μπορεί να προσφερθούν για να ε, υπάρχει περισσότερο κεφάλαιο για την ποιότητα και την ποσότητα των θέσεων εργασίας και τι νομίζετε ότι μπορεί να προσφέρει το πρόγραμμα, το Ταμείο, για, την, για αλλαγή στο παραγωγικό μας μοντέλο, κάτι που είναι απαραίτητο σε πολλές χώρες. Όχι απλώς να διοικητευτούν χρήματα σε προσωρινά προγράμματα και σε χώρες που ήδη τα πάνε καλά και δεν είχαν προβλήματα μέχρι τώρα σε αυτό το κλάδο. Ευχαριστούμε κύριε Τόρες που ήρθατε να μας μιλήσετε σήμερα το πρωί. Εγώ ήθελα να επιμείνω στα ίδια τα προγράμματα και την φύση τους, το χαρακτήρα τους. Μας τα εξηγήσατε καλά και συμφωνώ μαζί σας ότι τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να είναι νέα που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί από άλλες πηγές και προγράμματα σε νέους τομείς, τομείς προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ψηφιακή ε, τεχνολογία και ενέργεια. Όταν λέμε νέους τομείς, εννοούμε και νέες αρμοδιότητες βέβαια. Οπότε η ερώτησή μου είναι, οι άνεργοι, αυτοί που ψάχνουν δουλειά και μάλιστα αυτοί που ε, ψάχνουν από πολύ καιρό, γιατί όπως τα ξέρετε όσο περισσότερο καιρό αναζητά κανείς εργασία τόσο πιο δύσκολο είναι να επιστρέψει και στην αγορά εργασίας. Αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν ε, σύντομα θα υπάρχουν απαραίτητε δεξιότητες. Η πρώτη πρώτη επένδυση δεν θα πρέπει να είναι η δημιουργία και η προσφορά νέων δεξιοτήτων. Ευχαριστούμε για τα Στάινρουκ. Μετά τις ε, δηλώσεις σας μου ήρθε μια σκέψη χωρίς να την έχω εξετάσει τεχνικά. Τίθεται το ερώτημα μια που τα κονδύλια της πρωτοβουλίας για τους νέους δεν απορροφήθηκαν καθόλου από τα κράτη-μέλη. Μήπως έχετε σκεφτεί να χρησιμοποιήσετε αυτά τα κονδύλια ως μέρος του σχεδίου επενδύσεων για να προωθήσετε πολύ την ε, απασχόληση των νέων στην Ευρώπη. Τώρα έτσι μου ήρθε. Αλλά αφού χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις και θέλουμε ακριβώς να στοχεύσουμε τους νέους. Μήπως ε, είναι αυτό μια ευκαιρία. Η τελευταία ερώτηση από την κυρία τον κύριο. Από τον κύριο Φαν Ντενκελερε. Εάν θέλετε για να δώσουμε μετά το λόγο στον κύριο Τόρες και να μας απαντήσει. Ο κύριος Φάντον Κέντελερ. Ε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα παρατήρηση και παρουσίαση. Ως ε, ο νεότερος εδώ πέρα στην Επιτροπή σκέφτομαι ιδιαίτερα τους συνομιλίκους μου στην Ευρώπη και πραγματικά υπάρχει εδώ πέρα μεγάλη δυνατότητα δημιουργίας ε, θέσεων εργασίας ειδικά εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, αλλά το ζήτημα είναι πώς το συμφιλιώνουμε αυτό με την ανάγκη επενδυτών από ολόκληρη την Ευρώπη για το έργο του Ζακλου Γιούγκερ. Πώς ε, θεωρείτε ότι θα τους προσελκύσουμε, ειδικά στην Νότια Ευρώπη που πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Θεωρώ πως η ιδιώτες επενδυτές ε, θα θέλουν απόδοση στην επένδυσή τους. Κύριε Μπέκερ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια σύντομη ερώτηση. Γνωρίζετε εάν υπάρχει ένας τομέας αν γνωρίζετε τον τομέα ο οποίος από την αρχή της κρίσης ε, έχει σταθερή ανάπτυξη, η κοινωνική επιχειρηματικότητα. Ε, ξέρετε λοιπόν εάν η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελεί στόχο των επενδύσεων αυτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση ο κύριος Μάν. Ευχαριστώ. Έκανα και μία ερώτηση πριν, αλλά τώρα να επαναλάβω κάτι το οποίο είναι σημαντικό υπάρχει η δυνατότητα ε, και πρέπει βεβαίω να είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε δουλειές με προοπτική, με μια κατάρτιση. Θεωρείται λοιπόν πράγματα όπως η διπλή κατάρτιση που υπάρχει σε κάποια κράτη-μέλη θα πρέπει να προωθηθεί γιατί κάποια κράτη-μέλη λένε ναι, το θέλουμε. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να στηρίξουμε κάτι τέτοιο το οποίο έχει αποδειχθεί επιτυχημένο. Νομίζω πως έτσι θα έχουμε επιτυχία και με τους επενδυτές σε πολλά κρατημέλη. Μπορείτε να δώσετε μια σύντομη απάντηση σε όλες αυτές τις ερωτήσεις παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ και πάλι για την συναρπαστική συζήτηση. Νομίζω είναι σαφές πως πρέπει να συνεχίσουν αυτές οι συζητήσεις θα απαντήσω κατά ενότητες για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που αναφέρθηκε από πολλούς και αναφέρθηκαν και τα κριτήρια. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι δημόσια τράπεζα. Είναι φυσικό λοιπόν πως τα κίνητρα της πρέπει να είναι διαφορετικά, γιατί δεν χρειάζεται μια δημόσια τράπεζα για να παίξει ρόλο ενδιάμεσου που θα μπορούσε να το κάνει μια ιδιωτική. Το βασικό λοιπόν εδώ πέρα είναι να διασφαλίσουμε οπωσδήποτε ένα επίπεδο λειτουργίας και κερδοφορίας που θα είναι επαρκές, αλλά να δεχτούμε πως κάποια, αν όχι τα περισσότερα από τα ωφέλη του επενδυτικού αυτού σχεδίου θα πάνε στις ευρωπαϊκές χώρες στο σύνολό τους. Θα είναι αν θέλετε ένα κοινωνικό μέρισμα και η ιδιωτική, το ιδιωτικό κέρδος για την τράπεζα θα είναι πολύ μικρότερο. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζονται οι δημόσιες ε, τράπεζες, για να επενδύσουν ε, σε τομείς όπου το κέρδος το συλλογικό θα είναι πολύ μικρότερο από το ιδιωτικό. Αλλιώς θα κάνει και μια ιδιωτική τράπεζα. Οπότε το να δεχτούμε αυτά τα νέα κριτήρια για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όχι μόνο την κερδοφορία, αλλά για τον αντίκτυπο που έχει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Περιλαμβανομένων βεβαίω και των επενδύσεων. Ε, απαιτείται λοιπόν μια αλλαγή, για... τώρα δεν ξέρω εγώ ποια είναι γιατί δεν είμαι στην τράπεζα, των κριτηρίων για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Έγιναν πολλές ερωτήσεις για την ποιότητα των θέσεων εργασίας και την αξιοπρεπή δουλειά. Σημαντικές. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πράγμα που μπορεί να γίνει. Δηλαδή όταν έχουμε αυτά τα έργα για ψηφιακή οικονομία, ενέργεια, δίκτυα κτλ. Όταν γίνεται λοιπόν ένας διαγωνισμός για δημόσια έργα, εμείς έχουμε ένα μέσο για τις δημόσιες προμήθειες για να λαμβάνονται υπόψη ε, τα, οι προδιαγραφές ε, της εργατικής νομοθεσίας. Υπάρχει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά θα μπορούσε να γίνει μια πανευρωπαϊκή πολιτική έτσι ώστε να ε, υπάρχουν και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας επιπλέον. Στο σημείο 3 της έκθεσης θα ήταν κάπως υπερβολικό να ζητήσουμε από το έργο αυτό να ασχοληθεί με την ποιότητα των θέσεων εργασίας, αλλά είναι ένα πανευρωπαϊκό ζήτημα βεβαίως. Ε, κάθε έργο πρέπει να ασχολείται με αυτό. Και είναι καλύτερο για την απασχόληση να μπει το σχέδιο αυτό σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και στρατηγική απασχόλησης. Υπήρχαν επίσης ερωτήσεις για το ζήτημα της ε, νεολαίας και πώς θα εμπλακεί και των δεξιοτήτων. Θα υπάρχει νομίζω ένα στοιχείο εξορισμού που υπάρχει σε κάθε χώρα. Παράδειγμα της χάρη. Σε κάποιες χώρες οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν ήδη ε, πρόσβαση στις ε, τράπεζες. Αλλά δεν ισχύει αυτό σε όλες τις χώρες. Ανεργία υπάρχει γιατί σε πολλές χώρες υπάρχουν κερδοφόρες μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό το σχέδιο για να γίνει κάτι το οποίο δεν υπάρχει σε κάποιες χώρες. Και έτσι θα μπορούσε να ξεκλειδώσει αυτό το δυναμικό που υπάρχει. Το θέμα των ε, δεξιοτήτων. Καταλαβαίνω και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ε, Ίσως το έχουμε υποτιμήσει στην έκθεση, μπορούμε να το σκεφτούμε. Το αιώνιο ερώτημα είναι ποιες δεξιότητες. Είναι δύσκολο να το κρίνουμε απριόρι. Σημαντικό είναι να υπάρχει μια κάποιοι, να υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι θα μπορούν να ανοιχνεύουν γρήγορα ποιες είναι οι δεξιότητες που απαιτούνται για να αντιδρά το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Γιατί νομίζω είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψουμε το Υπάρχει μία περίοδος γρήγορης ε, τεχνολογικής αλλαγής με απρόβλεπτες συνέπειες. Κάποιοι άνθρωποι θεωρούν πως ε, δουλειές ρουτίνας ε, που απαιτούν και υψηλή εκπαίδευση θα φθήνουν τα επόμενα χρόνια. Και εξαρτάται τώρα, αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα μέρο σχεδίου ανάλογα με την χώρα. Τέλο, υπήρχε μια πάρα πολύ σημαντική ερώτηση για το γεωγραφικό στοιχείο του, του σχεδίου. Θα απαντήσω στα γαλλικά. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια ερώτηση κατά κάποιο τρόπο να εξετάσει δηλαδή κανεί σε ποιο μέτρο το επενδυτικό σχέδιο θα αποτελέσει το έμβριο μια ευρύτερης ευρωπαϊκής πολιτικής και ιδίως με το κοινό νόμισμα στη ζώνη ευρώ, όπου υπήρχε ένα ε, στοιχείο που ήταν ενεπαρκές, δηλαδή μια, πολιτική, μια οικονομική πολιτική. Εν τέλει θα χρειαστεί δηλαδή μια οικονομική πολιτική για να συμπληρώσει την νομισματική πολιτική. Μπορεί εδώ αυτό να, αποδειχθεί το έμβριο. Και το γεωγραφικό στοιχείο παρεμβαίνει εδώ για το 1 τρίτο του 1 εκατομμυρίου απασχολήσεων. Θεώσεων απασχολήσει δηλαδή για να ωφεληθούν οι περιφέρειες όπου έχουν λιγότερη απασχόληση τώρα. Αυτό λοιπόν το στοιχείο του εμβρίου. Είμαι βέβαιος ότι κάποιες ερωτήσεις θα έμειναν αναπάντητες, αλλά σας ευχαριστώ πολύ για την ε, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και για την ευκαιρία που μου δώσατε να εμφανιστώ σήμερα ενώπιον σας. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τόρες και είμαι βεβαία ότι θα θέλουμε να σας προσκαλέσουμε ξανά στην Επιτροπή μας κάποια στιγμή στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις διαφωτιστικές απαντήσεις που δώσατε. Ευχαριστώ και πάλι. Και τώρα θα ψηφίσουμε. Δώστε μας όμως ένα ή δύο λεπτά ε, να βρούμε τις κάρτες μας και ούτω καθεξής.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 Θα αρχίσουμε πάλι, λέει η Πρόεδρος, με τις ε, ψηφοφορίες ε, για, το, για τις ε, αιτήσει κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Παγκοσμιοποίησης. Αρχίζει η ψηφοφορία, η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Υπάρχουν τέσσερις πλεονάζοντες από το ΕΛΚ. Σας θέλουμε, αλλά... Εντάξει τώρα. Ωραία. Βλέπετε το αποτέλεσμα. Πέρασε τη Επόμενο. Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Βέλγιο, Σέντο κομπά, άρχεται η ψηφοφορία. Όντω ξεκίνησε. Πέρας. Εγκρίνεται. Αλλιώς Λάρα από τη Γερμανία. λόγος στη Γιώτα Ευχαριστώ. Η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών έχει υποβάλει μια προφορική τροπολογία για αντικατάσταση της παραγράφου 6. Εμείς δηλαδή προτείνουμε η παράγραφος 6 να αντικατασταθεί ως εξή και το λέω στα αγγλικά. Σημειώνει ως εκ τούτου ότι δεν προβλέπονται έξτρα κίνητρα για εκπαίδευση από το Ταμείο, πιο προσωποποιημένα μέτρα, ωστόσο, δηλαδή πιο εξειδικευμένα μέτρα θα πρέπει να ε, ενισχυθούν, να ενθαρρυνθούν. Μάλιστα. Οπότε θα ψηφίσουμε το σύνολο του κειμένου που τροποποιήθηκε προφορικό. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα απαλλαγή του Γενικού Προπολογισμού. Συμβαστική Α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται.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 υπέρ, κατά, πέρας της Εγκρίνεται. επτά υπέρ, κατά, αποσές, απορρίπτεται. οκτώ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9. Αποσύρεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Σ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19. Με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο της πρότασης όπως τροποποιήθηκε. Το σχεδίο γνωμοδότησης. Άρχεται ψηφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Απαλλαγή. Συμβαστική Α. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ. Ναι, υπάρχει και προφορική τροπολογία όπως βλέπετε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4. Παράγραφος 4 δεν θα ψηφιστεί. Οπότε ψηφίζουμε το σχέδιο γνωμοδότηση όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. απαλλαγή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4, παράγραφος 4, τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 5, τροπολογία 3. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Σχέδιο γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε, ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας. Εγκρίνεται. Σχέδιο γνωμοδότησης Ευρωπαϊκό, Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας. Δημοσιονομικό έτος 2013. Παράγραφος 2. Υπέρ. Με συγχωρείτε, τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Αγκρίνεται. 2. Υπάρχει και προφορική τροπολογία από τον ίδιο τον συγγητή την εισηγήτρια μάλλον, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρία, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τέσσερα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σχέδιο γνωμοδότησης ως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Σχέδιο γνωμοδότησης για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Τροπολογία Α. Συμβαστική α. Άρχεται η ψηφορία. Συμβαστική α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ναι, όχι, δύο. Της εισηγήτριας. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το, το σχέδιο νομοδότησης ω τροποποιήθηκε. Πέρα. Εγκρίνεται. Και σχέδιο έκθεση σχέδιο γνωμοδότηση μάλλον. για τους οργανισμούς κατά το δημοσιονομικό έτος 2013. Τροπολογία 1 του κυρίου Πυρίνσκι. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική α. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική β. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε για το σχέδιο γνωμοδότησης ως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Αγκρίνεται. Αυτά ήτανε. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό το τόσο ωραίο αποτέλεσμα. Ε, Στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Να πω λίγα λόγια. Πρώτα, η επί της εσωτερικής διαδικασίας. Είχαμε πάρα πολλές ε, συνεδριάσεις, ε, οι πρόεδροι των επιτροπών για την κατανομή των αρμοδιοτήτων. Και βεβαίως κάθε φορά τόνιζα την σημασία της Επιτροπής Απασχόλησης και το ότι βεβαίως πρέπει να παρακολουθεί το θέμα στενά. Βεβαίως τεχνικά η νομοθετική πρόταση έχει ελάχιστες κοινωνικές πτυχές. Όμως ο βασικός στόχος ε, είναι να δημιουργηθούν ακόμα καλύτερες δουλειές και να καταπολεμηθεί η ανεργία και ειδικά η ανεργία των νέων. Και δεν είναι ε, επενδύσεις ε, για τις ε, χρηματαγορές, είναι επενδύσεις για θέσεις εργασίας. Και βεβαίως αυτό είναι ένα πεδίο εμπειρίας της Επιτροπής μας. Οπότε ζήτησα να εμπλακεί η Επιτροπή μας ε, με βάση το άρθρο 54 του κανονισμού. Όμως ε, η διάσκεψη των Πρόεδρων των Επιτροπών ε, δεν έλαβε κάποια απόφαση παρά μόνο μία σύσταση για μία Επιτροπή η οποία θα συντονίζει και στην οποία θα συμμετέχουν όλες οι Επιτροπές του Κοινοβουλίου. Οπότε τώρα θα πρέπει να περάσουμε στην τελική κατανομή των αρμοδιοτήτων και είναι ε, πιθανόν η έκον να είναι η ε, αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή. Οπότε με ενημέρωσε η πρόεδρος ε, πως λόγω της ε, γρήγορης διαδικασίας κατά πάσα πιθανότητα δεν θα καταφέρουν ταυτόχρονα να προχωρήσουν σε μια πρωτοβουλία για σε μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για τα ζητήματα αυτά του ε, Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει το άρθρο 54 του κανονισμού και ορίσαμε την κυρία Βάνερ από τους Πράσινους και ξεκαθάρισα πολλές φορές και στους προέδρους των Επιτροπών και στον πρόεδρο της ΕΚΟΝ πως η Επιτροπή Απασχόλησης θέλει οπωσδήποτε η έκθεση αυτή της πρωτοβουλίας να γίνει εκ παραλλήλου με την νομοθετική πρόταση για να προωθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες από τις προτεραιότητές μας. Όμως δυστυχώς κάτι τέτοιο φαίνεται πλέον απίθανο, αλλά ακόμα θα το δούμε. Η ΕΚΟΝ όμως είναι επί αρμόδια όπως είπαμε. Οπότε πιθανό είναι η ΕΚΟΝ να είναι η επιστουσίας αρμόδια επιτροπή και οι υπόλοιπε επιτροπές να συμμετέχουν σε μια επιτροπή που θα κατευθύνει τις εργασίες και ακόμα και αυτό δεν είναι σίγουρο. Θα πληροφορηθώ και θα σας ενημερώσω το στομότερο δυνατόν. Έχουμε λοιπόν την πρώτη ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή μας για το ταμείο αυτό και θα δώσω τον λόγο στους ε, συντονιστές. Δεν βλέπω πως δεν υπάρχει όμως κανείς εδώ πέρα. Δεν ξέρω, κυρία Σαρτιέ μπορεί να μιλήσει εξ ονόματος του ΕΛΚ. Oh, sorry. But I don't have that. Sorry, I you. put it. I apologize. It's... my... Α, με συγχωρείτε. Η κυρία Γιασλοβιέσκα είναι ε, αρμόδια και θα πάρει το λόγο. Έχετε το λόγο. Ναι. Ναι, ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για, το, για την εμπλοκή σας και την προσπάθειά σας να αποκτήσει η Επιτροπή μας έναν ε, ισχυρότερο ρόλο στο θέμα αυτό. Επίσης ενδιαφέρουσα και η συνάντηση με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εργασίας. Η έκθεση αυτή έχει μεγάλη σχέση και με την έκθεση που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή για το κανονισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Σε αυτό το έγγραφο χιλιάδες Ευρωπαίοι βλέπουν μια ελπίδα για την βελτίωση της ζωής τους σε αυτούς τους καιρούς κρίσης. Θέλουμε να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία αλλά βλέπουμε πως ε, τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας ε, δεν επαρκούν. Υποτίθεται ότι θα ήταν ε, μια κινητήριος δύναμη για να ξαναξεκινήσει η οικονομία και θα έχει τρεις πυλώνες. Πρώτος είναι η χρήση 350 δισεκατομμυρίων ευρώ τα επόμενα τρία χρόνια έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των δημοσίων κονδυλίων και να πάρουν μπρος και οι ιδιωτικέ επενδύσεις. Ο δεύτερος πυλώνας είναι να φροντίσουμε οι επενδύσεις αυτές να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και ο τρίτος πυλώνας είναι η μείωση της γραφειοκρατίας για να γίνει η Ευρώπη πιο ελκυστική για επενδύσεις και να υπάρξει ένας ε, πολλαπλασιαστής για το ε, σχέδιο αυτό θα υπάρξει ένας πολυπρασιαστής όταν ενταχθούν στο Ταμείο περισσότερα κράτη-μέλη, αναπτυξιακές τράπεζες και ιδιώτες επενδυτές όπως ήδη τονίστηκε πολλές φορές. Το Ταμείο θα πρέπει να αποδείται για περισσότερες ιδιωτικές ε, επενδύσεις ε, παρά λοιπόν το ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το έγγραφο δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στην διάθεσή μας, άρα πρέπει να δράσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Πρώτα απ' όλα ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ ε, παρουσίασε το επενδυτικό σχέδιο πάρα πολύ γρήγορα στις 26 Νοεμβρίου πέρσι. Επίσης το Συμβούλιο ενέκρινε γρήγορα το σχέδιο στις 18 Δεκεμβρίου και ζήτησε από τους συνομοθέτες να ολοκληρώσουν τη δουλειά μέχρι το τέλος Μαρτίου. Ο Επίτροπος Ντομπρόφσκης επίσης τονίζει πως η ολοκλήρωση της εργασίας αυτής ε, είναι δυνατή λόγω της στήριξης που υπάρχει στο Συμβούλιο. Από όσο ξέρω, η Επιτροπή μας θα πρέπει να ψηφίσει τη γνωμοδότηση μέχρι τις 24 Μαρτίου. Έχουμε άρα δύο μήνες να αναπτύξουμε μια ισχυρή και συνεκτική θέση. Ε, εκτός ε, αν προκύψει κάτι λοιπόν, εκτός απροόπτου, θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες μας μέχρι το τέλος Μαρτίου, κάτι το οποίο σημαίνει πως το Ταμείο θα λειτουργεί ήδη στα μέσα του έτους. Πολύ γρήγορα λοιπόν. Σήμερα λοιπόν δεν θα συζητήσουμε συγκεκριμένες τροπολογίες, αλλά βεβαίως θέλουμε να ακούσουμε τις πρώτες σας εντυπώσεις και το πώς θα γίνει ένα ρεαλιστικό εργαλείο προώθησης της οικονομίας μας το ταμείο αυτό, πώς θα προωθήσουμε δηλαδή την Ατζέντα Ευρώπη 2020. Πριν παρουσιάσω όμως την δική μου προκαταρκτική θέση, να τονίσω πως 7 επιτροπές θα παρουσιάσουν τις γνωμοδοτήσεις τους ε, στην ε, έκθεση. Καμία από τις 7 επιτροπές αυτές δεν θα ασχοληθεί πολύ με τις κοινωνικές πτυχές, οπότε θέλω να το κάνει αυτό η δικιά μας επιτροπή. Όλοι γνωρίζουμε πως οι κοινωνικές πτυχές έχουν μεγάλη σημασία για την επιτυχία του Ταμείου. το έλλειμμα των επενδύσεων απειλεί τους στόχους της Ατζέντα 2020. Οι δράσεις οι οποίες αναλήφθησαν δεν έχουν οδηγήσει στα αναμενόμενα αποτελέσματα και έτσι θεωρούμε με βάση τα δεδομένα τα τωρινά ότι θα εξοδευτούν σωστά τα χρήματα αυτά στις μεταφορές, τα δίκτυα ενέργειας, την υποστήριξη της καινοτομίας. Ε, οι επενδύσεις λοιπόν θα στοχευθούν και θα στραφούν προς την πραγματική οικονομία και αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό του Ταμείου. Ε, τα έργα θα επιλεγούν με βάση την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία και το πόσο συμμορφώνονται με τους στόχους της πολιτικής μας. Ε, τέτοιες επενδύσεις θα πρέπει να μεταφραστούν σε δημιουργία θέσεων όσο το δυνατόν πιο μονίμων και υψηλής ποιότητας. Αλλά βεβαίως θα πρέπει να στηρίξουμε και διασυνοριακά έργα στο μέτρο του δυνατού. Διάφοροι ειδικοί λένε πως μπορούν να δημιουργηθούν μέχρι και 2,5 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. Η έρευνα δείχνει πως από σήμερα οι Ευρωπαίοι και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν πολλά εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Η ρευστότητα είναι αρκετά υψηλή. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων λέει πως αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε τώρα στην Ευρώπη είναι πως σημαντικά έργα και επικερδοί δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Όπως είπε ο Επιτροπός Κατάινεν, έχουμε μια κρίση εμπιστοσύνης η οποία δεν μας επιτρέπει να ε, υπάρξει μια επανεκκίνηση στην οικονομία. Επιπλέον, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18 19 σεπτεμβριου οι συνεισφορές ε, στο Ταμείο δεν πρέπει να επιβαρύνουν ε, τους υπολογισμούς του χρέους των κρατών μελών. Άρα θα πρέπει να αναπτυχθεί μια μεθοδολογία έτσι ώστε οι συνεισφορές ε, των κρατών μελών να είναι ουδέτερες ε, δημοσιονομικά. Επίσης, ε, έχω ήδη εκφράσει τις επιφυλάξεις μου για την χρήση του Ταμείου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να χρηματοδοτήσει διασυνοριακές επενδύσεις που θα οδηγήσουν σε περισσότερη ανάπτυξη και θα είναι στοχευμένα τα κονδύλια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, το Ταμείο θα χρησιμοποιήσει τα κονδύλια τα οποία δεν είχαν χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής. Ένα ερώτημα λοιπόν είναι το εάν υπάρχουν αρκετά τέτοια κονδύλια χρησιμοποιητά που θα χρησιμοποιηθούν τώρα. Έχουμε αρκετές εγγυήσεις ε, για να, ότι θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα κονδύλια μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν είμαι σίγουρη για το αν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να ε, κάνουν τόσα έργα. Πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί αυτές δημιουργούν θέσεις εργασίας. Επίσης, σημαντικό είναι να αναλύσουμε το εάν ο κανονισμός αυτός θα χρησιμοποιηθεί για να χρησιμοποιηθούν τα, τα, μία, τα κονδύλια του ΕΤΣΕ. Να δούμε δηλαδή επίσης αν θα δημιουργηθεί τελικά να δημιουργηθούν κάποιες συνέργειες. Οι αποφάσεις λοιπόν δεν πρέπει να βασίζονται σε πολιτικά κριτήρια. Αντιθέτως, τα έργα πρέπει να επιλέγονται με βάση επιχειρηματικά κριτήρια και την κερδοφορία. Εάν η συμμετοχή στην ε, Διευθυντική αυτή Επιτροπή βασίζεται στη συνεισφορά των κρατών μελών, τότε προφανώς τα κράτη-μέλη που δίνουν περισσότερα θα παίξουν το βασικό ρόλο και θα κάνουν κουμάντο. Εντάξει, κατανοητό από τη μία, αλλά πολιτικά κάπως ε, επίμαχο κάτι τέτοιο. Πρέπει να δούμε επίσης ήδη από τώρα τα κριτήρια επιλογής έτσι ώστε οι δυνητικοί επενδυτές να ξέρουν το εάν θέλουν να εμπλακούν ή όχι. Ε, κάτι άλλο σημαντικό είναι πως πρέπει να βρούμε καλούς διαχειριστές που θα επιλέξουν τα έργα και ειδικά τα επενδυτικά έργα. Ήδη Είχαμε μια δυναμική συζήτηση σήμερα το πρωί. Δεν θέλω τώρα να μακρηγορήσω άλλο. Αναμένω λοιπόν τις ερωτήσεις σας, τις γνώμες σας, αναμένω τη συνεργασία με την Επιτροπή και ολόκληρο το Κοινοβουλίο. Σας ευχαριστώ. Η Μαρία Ζωάου Ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τη συντονιστριά μας για αυτήν την παρουσίαση και καταρχάς να ευχαριστήσω για τις πληροφορίες που εσείς Πρόεδρε μας παρέσχατε για το πώς θα ενισχυθεί η επίδραση της Επιτροπής Απασχόλησης σε αυτή τη σειρά πρωτοβουλειών που έχουν αναλυφθεί. Είμαι στο πλευρό σας και συμφωνώ όταν λέτε ότι η έκθεση ιδίας πρωτοβουλία για, για το επενδυτικό πρόγραμμα πρέπει να συνταχθεί βάσει του άρθρου 54 ε, από την ε, πλευρά της νομικής βάσης. Όπως λέτε, η απασχόληση και υψηλή ποιότητας απασχόλησης είναι ο βασικός στόχος όλου αυτού του επενδυτικού προγράμματος. Τώρα, όταν μιλάμε για απορρίθμιση και για το στατηγικό ταμείο, καταλαβαίνουμε ότι αυτό βρίσκεται στα χέρια της διάσκεψης των Προέδρων. Θα δούμε λοιπόν ποια θα είναι η τελική του απόφαση. Όμως, εν τέλει, πρέπει να διοργανώσουμε τι δικέ μα εργασίε κατά τρόπον, ώστε να δώσουμε συγκεκριμένη μορφή, το δικό μας αποτύπωμα στην τελική μορφή του κανονισμού. Άκουσα την συνάδελφο του ΕΛΚ και να τονίσω κάποιες από τις δικές μας μέρημνες από την πλευρά των σοσιαλιστών και δημοκρατών. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι αυτό το νέο στρατηγικό ταμείο θα δημιουργήσει ε, καλής ποιότητας θέσεις απασχόλησης και ότι αυτό θα είναι ο βασικός του στόχος. Για αυτό το λόγο νομίζω ότι ένα σημείο όπου θα πρέπει να πιέσουμε αρχικά ιδιαίτερα είναι τα, κριτήρια επιλογής των προγραμμάτων των σχεδίων για να είμαστε βέβαιοι ότι τα κριτήρια αυτά δεν θα εξασφαλίζουν απλώς κερδοφορία αλλά οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές προτεραιότητες που έχουμε κατά νου και η δυνατότητα να δημιουργήσουμε καλύτερες θέσεις απασχόλησης θα ληφθούν υπόψη. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα κριτήρια την επιλογή των προγραμμάτων. Δεύτερον, όπως θα βλέπετε στον κανονισμό αυτό θα υπάρχει ένας διάβλος, ένας διάβλος για να εντοπίσουμε τα ενδιαφέροντα προγράμματα. Ε, σε αυτόν τον διάβλο θα συγκεντρωθούν εμπειρογνώμονες για να υποστηρίξουν τα κράτη-μέλη στον εντοπισμό των κατάλληλων προγραμμάτων. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι εμπειρογνώμονες που θα συμμετάσχουν θα λάβουν υπόψη τα κριτήρια πρόθεσης ε, των ε, καλών θέσεων απασχόλησης για την Ευρώπη. Όχι μόνο βάσει του κλασικού κριτηρίου της κερδοφορίας, του κέρδους. Έπειτα ένα κρίσιμο σημείο για το μοντέλο δίκησης, ε, διακυβέρνησης του Ταμείου. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η συμμετοχή θα έχουν στο στρατηγικό ταμείο όλα τα κρατημέλη. Γι' αυτό είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως υποσχέθηκε, να βεβαιώσει ότι στο κεφάλαιο του ταμείου, του ταμείου ε, η συμμετοχή στο κεφάλαιο του Ταμείου δεν θα ληφθεί υπόψη για την αποτίμηση της δημοσιονομικής ισορροπίας των κρατών. Υπάρχει όμως ένα σημείο όπου έχουμε μια ιδιαίτερη ανησυχία. Ε, αφορά τη συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων. Διότι εδώ η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνει μια διάκριση μεταξύ των κρατών μελών. μεταξύ όσων βρίσκονται στο προκλητικό ε, μέρος του Συμφώνου Ανάπτυξης και Σταθερότητας. Είναι βέβαιοι ότι στη δημοσιονομική τους αξιολόγηση δεν θα μετρήσει η συνεισφορά τους. Αλλά τα κράτη-μέλη που ακόμα βρίσκονται στο διορθωτικό τμήμα του Συμφώνου και είναι αρκετά αυτά τα κράτη-μέλη, θα πρέπει να καταβάλουν την προσπάθεια να περάσουν στη φάση της πρόληψης, αλλά θα πρέπει να τους επιτραπεί να έχουν στήριξη από το ταμείο, δηλαδή να τους επιτραπεί η συγχρηματοδότηση. Αυτό είναι ένα σοβαρό ε, θέμα διότι οι ανισότητες στις επενδυτικές ικανότητες των κρατών μελών θα διονυστούν αν δεν το αντιμετωπίσουμε. Το ίδιο και η ικανότητά τους να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Αυτές είναι οι βασικές μας ανησυχίες προς στιγμήν, αλλά θα συνεχίσουμε τη μελέτη του θέματος. Αυτά και ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο τον Ενρίκε Αλβεσόμπο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω ισπανικά. Περιμένω να βάλουν όλοι τα ακουστικά τους. Ε, έχουμε φτάσει στο κομμάτι της υλοποίησης, γι' αυτό θα προσπαθήσω να είμαι συνοπτικός και να περάσω στην ουσία. Δηλαδή, δεν θέλω να μιλήσω περί ιδεολογιών, διότι η δουλειά από τον κανονισμό αρχίζει τώρα. Θα το δούμε με λεπτομέρειες, θα υποβάλουμε ιδέες, αλλά αυτό που θα μας οδηγήσει είναι η πρακτική εφαρμογή. ό,τι έχει εγκρίνει το Κοινοβούλιο για να στηρίξει το πρόγραμμα του Κιούνκερ. Με μεγάλη χαρά διαπιστώνουμε ότι υπάρχει σύγκληση και πρέπει να συνεχίσουμε. Βεβαίω εδώ αντιδρούμε σε μια κατάσταση έκτακτη, ε, σε μια κρίση και γι' αυτό η Ευρώπη λαμβάνει μέτρα ε, και γι' αυτό θα πρέπει να παραμείνουμε και στα θέματα ουσίας. Υπάρχει μεγάλο δυναμικό για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Θα πρέπει λοιπόν να εξαλειφθούν οι φραγμοί και να επικρατήσουν οι κοινέ μα αξίε όπω η αξιοπρεπή εργασία και ούτω καθεξή. Όμω να μην ξεχνάμε ότι το πρόγραμμα Juncker ε, είναι ένα δις ευρώ που θα πολλαπλασιαστούν 1,4 από την ΕΤΕ και αυτό ελπίζουμε ότι θα ενισχυθεί και από, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ λοιπόν ε, πώς, ε, να προσέξουμε πάρα πολύ τι θα γίνει με αυτό το αρχικό κεφάλαιο των, ε, του 21 δισεκατομμυρίου των 21 θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα υπάρξει αυτή η μόχλευση για να φτάσουμε τα 300 δις και θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια σταδιακή προσέγγιση για να έχουμε δράσεις αποτελεσματικές ως προς την οικονομία, τις υποδομές που χρειάζονται στην Ευρώπη. Χρειάζονται επενδύσεις που να είναι αποδοτικές ως προς τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αυτή είναι η δική μας δουλειά. Υπ' αυτήν την έννοια θα φροντίσουμε να υποβάλουμε συγκεκριμένε προτάσεις. Επίσης θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως προς τα στοιχεία της ε, κενσιανής οικονομίας. Δηλαδή μας ενδιαφέρει να στηρίξουμε την ε, οικονομία στην πραγματικότητά της, όχι την ε, να επιδοτήσουμε. Μια παγίδα που την είδαμε πρόσφατα να προκαλεί προβλήματα. Ως προς το ρόλο της ΕΤ και για το Στατηγικό Ταμείο Επενδύσεων Έχουμε ξαναπεί εδώ ότι υπάρχει τεράστιο δυναμικό δημιουργία θέσεων απασχόληση με τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Θα δούμε πώ θα πάνε τα πράγματα, αλλά ο κανονισμό πρέπει να είναι ε, ένα πρακτικό εργαλείο και όχι ένα δόγμα. Ιδεολογικό. Σε κάθε περίπτωση η ουσία είναι να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης ποιότητας με σοβαρές διευθυντικές επενδύσεις. Είναι μετροπαθέ το πρόγραμμα Γιούνκερ, αλλά θα πρέπει όλοι να αποφελουθούν. Ευχαριστώ. Ζητήσατε το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχάς και εγώ να σας ε, συγχαρώ, όπως και οι συνάδελφοι, για τη συμμετοχή της Επιτροπής Απασχόλησης σε όλη αυτή την προσπάθεια. Είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε και την ε, παρουσία μας. Να μην ξεχνάμε το φόντο βέβαια όλης αυτής της πρότασης που είναι ότι δεν είναι πανάκια αυτή η πρόταση. Δεν θα αντιμετωπίσουμε συνολικά την ενεργεία, ούτε θα εξαλειφθεί η ενεργεία των νέων. Στην Ευρώπη υπάρχουν και διευθυντικά προβλήματα που συναντώνται σε όλες τις οικονομίες. Εδώ πρέπει να συγκεντρώσουμε τις προσπάθειές μας σε μια ανησυχία που μας έρχεται κατά νου συνέχεια όταν μιλάμε για το Στρατηγικό Ταμείο. Η Διευθύνουσα Επιτροπή, η Επιτροπή που θα επιλέγει τα διαφορετικά προγράμματα που συζητώνται, που θα έχουν υποβληθεί. Λένε ακούσαμε ότι θα είναι εξυπηρογνώμονε που έχουν εργαστεί στην αγορά. Δηλαδή θα δίνουν έμφαση στην αγορά και θα έχουν μαζί του και τα κομπιουτεράκια του για να υπολογίζουν τα αποτελέσματα. Νομίζω και οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να συμμετάσχουν. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες. Να μην δοθεί έμφαση μόνο στην αγορά και τις ανάγκες της, αλλά και στην απασχόληση. Θα πρέπει να δούμε τον αριθμό των θέσεων που θέλουμε να δημιουργήσουμε, αλλά να μην είναι θέσεις ε, από άχυρο που να τις πάρει ο αέρας πολύ γρήγορα να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει κόσμος που δουλεύει και τελικά δεν κερδίζει τίποτα. Αυτό ε, μας ενδιαφέρει. Πώς θα εξασφαλίσουμε παρουσία των ε, κοινωνικών εταίρων στην ε, Διευθυνής Επιτροπή και κάτι ακόμη. Πρέπει να καταλήξουμε σε μια θέση ε, ισχυρή. Δεν είναι τα κονδύλια αυτό που θα καθορίσει την βαρύτητά μας στο Ταμείο. Πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να μπορούν να συμμετάσχουν. Όλα. Και όλα θα έχουν να πούν την κουβέντα τους ως προς την ε, εφόσον υπάρχει δίκαιη συμμετοχή, αλλά το πιο σημαντικό είναι το είδος των θέσεων απασχόλησης που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Και πώς θα το κάνουμε αυτό. Να είναι ποιοτικέ θέσεις που από την αρχή της διαδικασίας να εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Ευχαριστούμε κυρία Βάνα. Μόνικα Βάνα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για την προσπάθεια που κάνατε, τη δέσμευση που κάνατε για να μεγαλώσει ο ρόλος της Επιτροπής Απασχολήσεως και που βρίσκω ότι είναι απόλυτα απαραίτητη. Γιατί όπως είπατε και εσείς αλλά και άλλοι, η δημιουργία απασχόλησης και η κοινωνική διάσταση του επενδυτικού σχεδίου για την επίτευξη των στόχων του 2020 είναι ένα ή ίσως και ή, ε, ένας από, ή και από πιο, πιο σημαντικούς στόχους. Θα πρέπει να είναι πιο σημαντικούς στόχους του επενδυτικού σχεδίου. Και νομίζω ότι η διάσταση αυτή δεν έχει ακόμα εξασφαλιστεί. Ως πράσινη θα θέλαμε, και το είπατε κι εσείς, ε, να γίνει εκ παραλίλου μια δουλειά για την έκθεση και για την πρόταση νομοθετικού περιεχομένου ψηφίσματος, γιατί είπατε και εσείς ότι χρειάζεται ένα ευρύ φάσμα για να περιληφθούν όλες οι απόψεις μας. Ήδη η συζήτηση που διεξάγεται τώρα, το έδειξε άλλωστε και ο ILO με την έκθεσή του, ότι δεν πρόκειται μονάχα για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αλλά και για το ποιόν των θέσεων αυτών απασχόληση που θα δημιουργηθούν, το πού, σε ποιε περιφέρειες θα δημιουργηθούν, ποια συνοδευτικά μέτρα θα ληφθούν ενεργό δηλαδή πολιτική απασχόληση και σε ποιου τομεί θα δημιουργηθεί η απασχόληση. Όλα αυτά πρέπει να επικαλύπτονται και με τη δική μας εργασία. Και όπως είπε και η ΑΕΛΟ, να μην υποφεληθούν μονάχα οι μεγάλοι όμιλοι επιχειρήσεων, αλλά τελικά και οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι. Το ερώτημα είναι τι πάει να πει καλή επένδυση σύμφωνα με την άποψη της δικής μας Επιτροπής Απασχόλησης. Άρα εδώ χρειάζονται quality jobs, καλές επενδύσεις σημαίνουν επενδύσεις που μειώνουν τη φτώχεια, μειώνουν τις ανισότητες και μας φέρουν κοντύτερα στους στόχους της Ευρώπης 2020. Χρειάζεται λοιπόν το κοινοφελέ στοιχείο, το κοινό καλό. Άκουσα τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Κατάινεν στην Επιτροπή Προϋπολογισμών να λέει ότι η βασική στόχη του σχεδίου επενδύσεων είναι η προσέλκυση επενδυτών και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Εμένα αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ λάθος προσέγγιση. Πιο πολύ πρέπει να μας ενδιαφέρουν οι επενδύσεις κοινοφελούς χαρακτήρα και ούτε μπορεί να είναι καθαρά επενδυτικό πακέτο υπέρ των επενδυτών. Πρέπει να ενισχύσει τις εργαζόμενες και τις φτωχότερες στον, ε, του ευρωπαϊκού ε, πληθυσμού. Κάτι το οποίο με ενοχλεί πολύ και το ακούω ξανά και ξανά και το λέω εγώ, το βλέπω σε ορισμένε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ, είναι ότι έχω την εντύπωση ότι με το σχέδιο επενδύσεων πάνε να φτιάξουν μια νέα δομή τη επενδυτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεχνώντας τις εμπειρίες που έχουμε συλλέξει από τις διάφορες δομές που έχουμε ήδη στην επενδυτική πολιτική, διότι έχουμε την πολιτική συνοχής, έχουμε τα διαφθορτικά ταμεία με μεγάλο όγκο επενδύσεων που ήδη έχουν καλή θετική στόχευση και καλή οργανωτική διαμόρφωση με δημοκρατικό χαρακτήρα άρα έχουν μια ξεκάθαρη δέσμευση υπέρ των στόχων της Ευρώπης 2020, άλλωστε λαμβάνουν καθαρά υπόψη και την περιφερειακή συνοχή, τους ε, τοπικούς περιφερειακούς φορείς, κοινωνικούς εταίρους, κοινωνία των πολιτών, όλα αυτά να ληφθούν υπόψη και όλα αυτοί να ενταχθούν μέσα στον σχεδιασμό των επενδύσεων. Το ίδιο να τονιστεί ο ρόλος των ε, δημοσίων υπηρεσιών, δηλαδή των κοινοφιλών ενώ υπηρεσιών. Όλα αυτά πρέπει να μπουν στο σχέδιο γιατί αλλιώς αν λησμονηθούν φτιάχνουμε πια μια παράλληλη δομή με τον κίνδυνο, το λέω κάπως υπερβολικά εδώ, οι φτωχές χώρες μέλη να αρκεστούν μοναχά στα διορθωτικά ταμεία και οι πλούσιες χώρες να έχουν το νέο επενδυτικό σχέδιο με άλλους κανόνες και εκεί βεβαίως θα ε, υπάρχει και δημοκρατικό έλλειμμα του steering board, αυτά όμως τα είπαν και άλλες ε, βουλευτές που μίλησαν πριν από μένα. Ε, να φανεί καθαρά λοιπόν ότι οι κατευθυντικές γραμμές των σχεδίων επενδύσεων του steering board και ούτε καθεξής είναι στοχευμένες υπέρ της επιλογής των έργων με δημοκρατική ευθύνη. Αυτό νομίζω είναι από τα πιο σημαντικά καθήκοντα που ε, έχουμε μπροστά μας ως Επιτροπή Απασχόλησης. Και είναι κατεπήγον να αρχίσουμε τώρα τη δουλειά μας. Θα συμφωνήσω με όλες τις άλλες βουλευτές που, μιλ, που τα είπαν αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από από το Λύκειο στα μαθήματα ελληνικού, ελληνικών και φυσικής μας έλεγε η καθηγήτρια μαθηματικών ότι ε, όταν ε, πηγαίνει κανείς σε ένα τέτοιο άγνωστο πεδίο είναι σαν να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα σε αυτοκινητόδρομο και αυτό το λέω γιατί τα μαθηματικά δεν ήταν το καλό μου μάθημα. Ε, για το στατηγικό λοιπόν ταμείο αναρωτιέμαι κατά πόσο είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε τα αριθμητικά στοιχεία που μας έχουν πετάξει. και εγώ αναρωτήθηκα ήδη αν πως το πρόβλημα ήταν αυτό το παλιό με τα μαθηματικά αλλά μάλλον καλά κατάλαβα όταν λέμε για ένα δις για το Ταμείο Στατηγικών Επενδύσεων αντιλαμβάνομαι ότι 6 θα έρθουν απευθείας από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέντε από την ΕΤΕ και τι θα πει αυτό. Ε, δεν ε, ε, επινοούμε κονδύλια, αλλά τα παίρνουμε από εκεί που είναι διαθέσιμα. Λόγω χάρη θα περικοπούν από την έρευνα που θα έπρεπε να είναι ακριβώς κινητήριο δύναμη που θα δώσει οξυγόνο στην οικονομία μας και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και ε, με αυτό το εφάνταστο πρόγραμμα ε, του Πρόεδρου Γιούγκερ παίρνουμε κονδύλια από προγράμματα όπως το ορίζοντας που ήδη λειτουργούν και τα διαθετεύουμε σε άλλα φαντασιακά προγράμματα. Επίσης διερωτήθηκα και το εξή. Αυτά τα κονδύλια έρχονται από ιδιώτες. Ε, για εξηγήστε μου, γιατί και εδώ δεν πολύ καταλαβαίνω, γιατί ε, από εδώ και μπρος οι ιδιώτες θα πρέπει να επενδύσουν σε αυτό το ταμείο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν εγγύησεις. Δεν υπάρχει εγγύηση. Ως τώρα οι ιδιώτες επενδυτές έχουν επιφυλαχθεί και δεν επενδύουν ε, ενώ ε, αντιθέτως ε, τώρα ξαφνικά θα βρούμε ένα εκατομμύριο επενδυτές που θα θέλουν να επενδύσουν. Ο Γιούνκερ επίσης είπε ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να συνεισφέρουν και να δώσουν κίνητρα για τη χρηματοδότηση αυτού του στρατηγικού ταμείου. Για να γίνει ελκυστική η πρότασή του, είπε ότι θα προβλέψει διευκολύνσεις για, την, για τον υπολογισμό του ελλείμματος στο ΕΠ. Ε, άριστα, όμως ξέρουμε ποια θα είναι η, η, ε, αντίδραση στις προτάσεις και τις υποβολές προγραμματών. Δεν είδα να γίνεται καμία νήξη για τον περιφερειακό χαρακτήρα των προγραμμάτων. Δηλαδή περιοχές δεν θα ευνοηθούν ως προς την επιλογή των προγραμμάτων. Όλα αυτά τα ε, κονδύλια θα μπουν στο ίδιο τσουβάλι και δεν θα υπάρχει καμία ε, διάκριση γεωγραφική. Δηλαδή η συνεισφορά της Ιταλίας μπορεί τελικά να χρηματοδοτήσει και να θυμίσω το παράδειγμα της Ιρλανδίας, αλλά δεν θέλω να παρεκτραπώ και να μακρηγορήσω, αλλά μπορεί να χρηματοδοτήσει προγράμματα και υποδομές άλλων χωρών. Ε, ποιο κράτος που έχει λίγο ε, μυαλό στο κεφάλι του, ένα κουκούτσι μυαλό στο κεφάλι του, θα ε, κάνει τέτοιες άμεσες επενδύσεις σε άλλα κράτη μέσω του εθνικού του προπολογισμού. Ας μιλήσουμε λίγο και για το χρονοδιάγραμμα, διότι προφανώς ε, ο χρόνος είναι πάρα πολύ απλωμένος στον ορίζοντα. Ε, ο Γιούνκερ είπε ότι το πρόγραμμα θα αρχίσει να λειτουργεί μέσα στο δεύτερο εξάμενο του 2015. Όμως αυτή είναι οι πρώτοι έξι μήνες που απαιτούνται για να δημιουργηθούν ε, οι διοικητικές δομές. Δηλαδή δημιουργούμε ένα νέο καινούριο δημιούργημα για αυτό το, για αυτό το νέο πρόγραμμα. Έπειτα διάφορες επιτροπές θα αποφασίζουν ποια προγράμματα πρέπει πρέπει να ε, χρηματοδοτηθούν. Για φανταστείτε πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να καταλάβει κανείς ε, ποιο είναι το χρησιμότερο πρόγραμμα, ποιο θα στηριχθεί και ποιο όχι. Και άλλοι μήνες που θα περάσουν έτσι. Με έναν χοντρικό υπολογισμό και θυμίζω ότι δεν είμαι καθόλου καλή στα μαθηματικά, αλλά σε έναν υπολογισμό έτσι κάπως ε, κατά προσέγγιση, θα έλεγα ότι από το πρώτο ευρώ που θα επενδυθεί σε αυτό το ταμείο θα φτάσουμε τουλάχιστον στο πρώτο εξάμεινο το 2016. Ξέρετε όμως πολύ καλά ποια είναι τα όρια του ταμείου. Θα έχουμε βγει εκτός χρονοδιαγράμματος ε, και χωρίς πρόβλημα και τι θα γίνει με, το, με τη μαγική μας ε, με το μαγικό μας ραβδί θα γίνει το Ταμείο Πενταετούς διά, Διάρκειας και ξέρουμε τι ε, φρικτά ναυάγια έχουν αυτά τα μακροπρόθεσμα, μακρόπουνα ε, σχέδια. Ενώ στην πραγματικότητα χρειαζόμαστε άμεσα προγράμματα με πρώτο θεμελιώδη σκοπό όχι να δημιουργήσουν απασχόληση, να λύσουν ένα μικρούλικο, ένα ελάχιστο πρόβλημα που ονομάζεται απόλυτη ένδυα. Διότι ακόμη σήμερα δεν καταλαβαίνουμε να κατανοήσουμε εάν τα στατιστικά στοιχεία έχουν λάβουν υπόψη ένα βασικότατο στοιχείο, όχι τον κίνδυνο ένδυας που διατρέχουν οι Ευρωπαίοι πολίτε, αλλά την απόλυτη φτώχεια, τι συνθήκε απόλυτη φτώχεια στην οποία ζουν πάρα πάρα πολλοί Ευρωπαίοι πολίτε να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης, αλλά ξεκινήσουμε ε, χωρίς να αφήνουμε νηστικά τα παιδιά που πεθαίνουν από δυσεντερία ή από ε, πείνα. Και μετά ας κάνουμε ό,τι επενδύσεις θέλουμε. Ευχαριστούμε Μαρία Αρενά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να συμβάλλουμε ω Επιτροπή Απασχόλησης όλη αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε στο βαθμό που η προβληματική που μας απασχολεί σήμερα είναι η απασχόληση στην Ευρώπη. Εάν υπάρχουν επενδύσεις θα πρέπει να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Θα συμφωνήσω με αυτό που είπε η συνάδελφο, η Μαρία Ζουάου για ό,τι αφορά την ε, ε, οργάνωση και τη λειτουργία του Ταμείου. Όμω να μιλήσω και για τα σχέδια στήριξη των προγραμμάτων. Μιλήσαμε για δείκτε που θα είναι δείκτε δημιουργία θέσεων απασχόληση, αλλά να είμαστε σίγουροι ότι οι μελέτε αντικτύπου για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση, να είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι μελέτε αντικτύπου ευρωπαϊκή κλίμακα. Ξέρουμε ότι ένα πρόγραμμα επενδύσεων σε μια συγκεκριμένη χώρα μπορεί να οδηγήσει σε μεταφορά θέσεων εργασία από τη μια χώρα στην άλλη. Να δούμε λοιπόν τον αντίκτυπο, να αναλύσουμε το τι θα προκαλέσει δημιουργία θέσεων απασχόληση με ένα τρόπο συνολικό, σφαιρικό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόγραμμα θα προσφέρει ε, θέσει απασχόληση ή απλώ θα μεταφέρει θέσει από τη μια χώρα στην άλλη. Το βρίσκω σημαντικό αυτό. Να το δούμε και έτσι. Το δεύτερο είναι είναι το θέμα της χρηματοδότησης. Εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λόγω χάρη σε συγκεκριμένους βιομηχανικούς τομείς, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η οι δεξιότητες των εργαζομένων μπορούν να συνδυαστούν με αυτούς τους βιομηχανικούς τομείς. Αυτή τη στιγμή βλέπω να υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ των δεξιότητων των εργαζομένων και ιδίω των νέων που φεύγουν από το σχολείο χωρίς να έχουν συγκεκριμένε δεξιότητε και την απόσταση που απαιτούν και την, ε, τις ανάγκες που ζητούν να καλύψουν οι νέοι τομείς της βιομηχανίας. Θέλουμε λοιπόν προγράμματα στήριξης των εργαζομένων που ενδεχομένως θα μπορούσαν να λάβουν αυτές τις νέες θέσεις εργασίας. Σήμερα βλέπουμε ότι αντιθέτως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής η τάση είναι να μειώνεται η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης ή η χρηματοδότηση της κατάρτισης, οπότε θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με, για αυτή την προσφορά και ζήτηση που θα δημιουργηθεί μέσω αυτών των προγραμμάτων. Τέλο, πολύ συχνά γίνεται λόγο για καινοτομία στα διάφορα προγράμματα. Η καινοτομία δεν ε, προκύπτει από τι νέες τεχνολογίες. Εάν μιλήσουμε για τα προγράμματα τεχνολογική μετάβαση ε, μετάβαση προ ε, θέσει απασχόληση υψηλών προσόντων. Σε αυτήν την ενεργειακή μετάβαση υπάρχουν και χαμηλών προσόντων θέσει, όπω στον τομέα το κατασκευαστικό. Εάν λοιπόν ένα κράτο μέλο θέλει να επενδύσει να κάνει κρατικές επενδύσεις. Για να βεβαιωθεί ότι τα κτίρια του δεν θα είναι ενεργοβόρα. Εδώ μπορούμε να έχουμε βιώσιμα προγράμματα και από την πλευρά της ενέργειας και της απασχόλησης και τέτοιες επενδύσεις κρατικές πρέπει να στηριχθούν ε, οπωσδήποτε για την ενεργειακή μετάβαση. Αυτή τη στιγμή ακούω πολύ λόγος να γίνεται για τις ιδιωτικές επενδύσεις, για κερδοφορία από οικονομικής ε, πλευράς. Νομίζω η κερδοφορία πρέπει να είναι και ε, περιβαλλοντικός και κοινωνικός κερδοφόρα. Και βιώσιμη. Ευχαριστούμε Τζέιν Κόλλινς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. 350 εκατομμύρια ευρώ ε, μας είπε ο κύριος Γιούγκερ θα επενδυθούν σε όλη την Ευρώπη με αυτό το πρόγραμμα. «315 δις λοιπόν θα επενδυθούν σε όλη την Ευρώπη, αλλά δεν φαίνεται να περισσεύουν σε κανέναν αυτά. Ε, τα κράτη-μέλη έχουν κάπως πτωχεύσει, έχουν ε, επιβάλει αυστηρά μέτρα λιτότητας λόγω της αποτυχίας του ευρώ. Ή των, της κακοδιαχείρισης της δικής τους της ίδιας της οικονομίας. Δεν καταλαβαίνω από πού θα προέλθουν αυτά τα κονδύλια. Έτσι, λίγο πολύ θα πρέπει να βρούμε με ένα μαγικό τρόπο αυτά τα 315 δις. Λέγεται ότι τα περισσότερα θα προέρθουν από ιδιώτες επενδυτές. Πώς θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα. 21 δις ε, για την εγγύηση του Ταμείου και μετά για κάθε ευρώ που θα δαπανάτε από την Ένωση ε, στο τμήμα του κινδύνου κάθε προγράμματος θα ε, αναλογούν 4 ευρώ επένδυσης από τον ιδιωτικό τομέα. Μετά ε, γίνεται ένας θολός υπολογισμός όπου πολλαπλασιάζονται τα 21 δις επί 15 και καταλήγουμε στο 315 δις. Όταν θέτουμε ερωτήσεις σχετικά μας λένε ότι βασιζόμαστε στην υπόθεση ότι αυτό έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Όλο αυτό το σύστημα βασίζεται σε πάρα πολύ εποπτούς υπολογισμούς. Είναι πολύ ασταθείς αυτές οι υποθέσεις και δεν καταλαβαίνουμε πώς θα λειτουργήσει αυτό με την ιδιωτική επένδυση. Και για να είμαι ειλικρινής, όπως όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα, η κοινή αγροτική πολιτική, η κοινή αληφτική πολιτική και να μην ξεχνάμε και το εγχείρημα του ευρώ. Όλα πνίγηκαν σε ευρωπαϊκά προγράμματα και οδηγήθηκαν σε καταστροφή. Το να γυρνάμε λοιπόν και να λέμε ότι 15 δις θα μας έρθουν από το πουθενά είναι μια πάρα πολύ ευσεβής επιθυμία και πόθος αλλά είναι μια παραπλανητική προσπάθεια να κερδίσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Οι εμπειρίες του Ηνωμένου Βασιλείου με τα μεγάλα δαπανηρά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησαν σε διοικητικό άχθος με χρήμα να μην πηγαίνει σε αυτούς που πραγματικά το χρειάζονταν με απάτη και διασπάθηση. Οι ευρωπαϊκοί ε, λογαριασμοί βέβαια δεν έχουν ε, εγκριθεί εδώ και δύο δεκαετίες. Ε, και το Ταμείο λέει ότι με 315 δις θα σώσει το ευρώ. Και δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Ακόμη όμως και αν το βρούμε αυτό το ποσό, δεν θα υπάρξει λύση. Διότι υπάρχουν χώρες που έχουν τελείως διαφορετικές, ριζοσπαστικά διαφορετικές οικονομίες εντός του ευρώ και οι οποίες είναι αλληλένδετες. Αυτό όμως έχει οδηγήσει στην καταστροφή την Ελλάδα, την Νότια Ευρώπη και εκατομμύρια ε, πολίτες που έχουν πληγήσει σε όλη την Ευρώπη. Ε, όσα χρήματα και αν ρίξει κανείς από τον κορβανά, δεν θα σωθεί η ε, ασθμένουσα, η ψυχοραγούσα αυτή ένωση. Thomas Mann. Thomas Mann. Μάλιστα. Η τελευταία παρατήρηση για στο Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Ακούστηκαν κάποια πράγματα τα οποία δεν ήταν πάρα πολύ σωστά. Η Ιταλίδα αδελφό στην εξάλεπτη ε, παρουσίασή της νομίζω ότι λέει κάποια πράγματα που ταιριάζουν περισσότερο σε προεκλογικό αγώνα ίσως. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι η ουσία εδώ πέρα. Πρέπει να πούμε πως έγινε μια νέα αρχή μέσω μιας νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ θέλει να θέσει διαφορετικές προτεραιότητες. Δεν θέλει μόνο να μιλήσει για την βιωσιμότητα των δημοσίων προγραμμάτων, αλλά χρειάζεται και μία εκτίμηση του κοινωνικού αντικτύπου, κάτι το οποίο βεβαίως πρέπει να συζητήσουμε και αυτό είναι καινούριο. Θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποκτήσει ένα κοινωνικό προφίλ. Σημαντικό αυτό. Οπότε το να λέμε ότι όλα αυτά δεν θα γίνουν και δεν σημαίνουν τίποτα δεν είναι και πολύ σωστό και υπεύθυνο. Αυτή η συζήτηση θα γίνει οπωσδήποτε και με την... Ε, και θα γίνει όπως ε, χρειάζεται. Δεν ξέρω αν έχουν συνειδητοποιήσει όλοι και όλα τα κράτη-μέλη πως έχουμε μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια νέα δομή, μπορούν να τεθούν διάφορα ζητήματα με δικαίωμα βέτο και τέτοια πράγματα, αλλά μιλάμε πάντα για ένα συλλογικό όργανο και με οποιαδήποτε προτεραιότητα να έχουμε, νέα ανταγωνιστικότητα, ανάπτυξη, αλλά βεβαίως ε, υπόψη να λαμβάνουμε και την κοινωνική πτυχή την απασχόληση δεν είναι κάποια νομεγκλατούρα όλο αυτό το ζήτημα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Ξέρω πως υπάρχουν μεγάλες διαφορές στα κράτη-μέλη. Εγώ μίλησα και είχα κάνει μια έκθεση για το ευρωπαϊκό πλαίσιο δεξιοτήτων, για την αμοιβαία αναγνώριση. Πρέπει λοιπόν να έχουμε συγκρίσιμες καταστάσεις έτσι ώστε να μπορεί να υπάρξει μια τέτοια ποιότητα και εκεί πέρα ακριβώς θα καταφέρουμε να προσελκύσουμε και τους ιδιώτες επενδυτές. Κάποιοι λένε πως δεν θα γίνει τίποτα και δεν θα έρθουν ούτως ή άλλως οι ιδιώτες επενδυτές. Μα άμα αισθανθούν πως υπάρχει ένα σίγουρο πλαίσιο και μπορούν να βασιστούν οι λογικοί επενδυτές θα έρθουν πιστεύω εγώ. Δεύτερη παρατήρηση. Λέτε πως τα νούμερα δεν βγαίνουν, τα 16 δισεκατομμύρια που έχουμε από τον προϋπολογισμό μας και τα 6 δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και υπάρχει μια μόχλευση. Εντάξει, μπορούμε να πούμε αν ισχύει αυτή η μόχλευση ή όχι και πώς θα φτάσουμε στα 300 τόσα. Έχουμε ιδιώτες επενδυτές που θέλουν και πρέπει να επενδύσουν σε σίγουρα έργα. Το ερώτημα λοιπόν είναι πότε ακριβώς θα εμπλακούν. Εάν μιλάμε για έργα που απασχολούν ανθρώπους, κατάρτιση κτλ. Ναι, αν υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις ε, έτσι ώστε να υποβάλει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σοβαρά και ξεκάθαρα έργα ή ε, να, και να μην είναι έργα τα οποία θα έχουν πάει τόσο χάλια σε εθνικό επίπεδο που θα πούν τα κράτη-μέλη ας τα δώσουμε στην Ευρώπη. Και να σταματήσουμε επιτέλους να κακολογούμε τα πάντα πριν καν ξεκινήσουν έτσι χωρίς την παραμικρή ευκαιρία. Εγώ χαίρομαι επίσης που έχουμε φιλόδοξο και γρήγορο χρονοδιάγραμμα. Αν είναι πάλι να περιμένουμε, πάλι να γίνονται όλες αυτές οι ατελείωτες συζητήσεις και να, λέμε, να κλαίμε τη μοίρα μας εδώ πέρα, δεν θα γίνει τίποτα για την ανεργία. Ε, οι άνθρωποι αυτοί έχουν δικαίωμα να δουν συγκεκριμένες αλλαγές και εδώ πέρα έχουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο, φιλόδοξο. Κυρία Πρόεδρε, σωστά είπατε θα πρέπει επιτέλους να ανταποκριθούμε και στον τίτλο μας που είναι Επιτροπή Απασχόλησης. Έχετε, Έχετε απόλυτο δίκιο. Απαντάει η Πρόεδρος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να λάβει το λόγο. όχι από ό,τι φαίνεται. Καλά λοιπόν. Α, μια στιγμή, η κυρία Αρταμεντιέρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όχι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τότε θα επανέλθουμε βεβαίως, έτσι, θα επανέλθουμε στο FC, θα επανέλθουμε ξανά και ξανά και βέβαια θα ενημερώσω και τους συντονιστές καθώς και την Ολομέλεια της Επιτροπής Απασχολήσεως για τις εξελίξεις. ώστε να μην λαμβάνετε πληροφορίες από αναξιόπιστες πηγές. Εσείς τώρα κύριε Γιασλοβιέτσκα, πέστε λίγα λόγια πριν να σας ε, ανακοινώσω το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Εγώ επιθυμώ να αναφερθώ σε ορισμένα σημαντικά σημεία που θα πρέπει να τα περιλάβουμε και στην υποβολή τροπολογιών. Η κυρία Ροντρίγκε μίλησε για τα κριτήρια επιλογής και άλλοι ή άλλε μιλήσατε για αυτά. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικά τα κριτήρια επιλογής και να λάβουν υπόψη το δυναμικό ή την δυνατότητα δημιούργησης απασχόλησης. Δημιουργίας, συγγνώμη, δημιουργίας απασχόλησης. Και όλες οι χώρες μέλη να μπορούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία διαχείρισης. Θα υπάρξει ενδιαφέρον από τις χώρες μέλη για τη συμμετοχή αυτή. Καλό είναι βέβαια να περιληφθεί το σχετικό στοιχείο. Το ίδιο για την συγχρηματοδότηση που επίσης είναι σημαντική υπόθεση να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ισότιμη πρόσβαση για όλες τις χώρες μέλη, ανεξάρτητα από την τρέχουσα κατάστασή τους και ίσως ιδίω για τις χώρες εκείνες που αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις. Να έχουμε δηλαδή, να περιλάβουμε κάποια στοιχεία που να τους το επιτρέψουν. Η κυρία Γκονζάλες έχει αποχωρήσει, αλλά ε, μίλησε για αυτό το θέμα. Να εξασφαλίσουμε ότι τα κριτήρια ευνοούν επενδυτικά έργα τα οποία θα επιτρέψουν δημιουργία απασχόλησης. Μιλούμε για δημιουργία 2,5 εκατομμυρίων θέσεων απασχόλησης. Γνωρίζουμε όμως ότι χρειαζόμαστε δεκάδες εκατομμυρίων θέσεις απασχόλησης για να αρχίσει πια να υπάρχει κάποια ασφάλεια στην αγορά εργασίας στην Ευρώπη. Η κυρία Κάρη μίλησε για την συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Μάλιστα, εγώ νομίζω ότι μπορούν να παίξουν ουσιαστικό ρόλο οι κοινωνικοί εταίροι. Δεν ξέρω εάν μπορούμε να εγγυηθούμε το ρόλο αυτό μέσα σε αυτό το νομοθέτημα. Αλλά θα πρέπει να αναζητήσουμε δυνατότητες ώστε να μπορέσει αυτό να γίνει. Αν θυμάστε χθε, στη διάρκεια της συζητήσεως, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κατάινεν είπε ότι θα υποβληθούν εκθέσεις. Εμείς βέβαια τις λαμβάνουμε αυτές μια φορά το χρόνο. Μπορούμε όμως να ζητούμε να υποβάλλονται εκθέσεις και να γίνονται αυτές μάλιστα και ανατρίμηνο έτσι ώστε να αποτελέσουν την βάση για το monitoring ε, από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σωστά είπε η κυρία Βέρνερ ότι έχουμε ήδη πολύ υλικό που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να θεσπίσουμε ε, ικανά κριτήρια. Για παράδειγμα έχουμε τα κριτήρια των διαρθρωτικών ταμείων που με κάποιο τρόπο εκπληρώνουν και το στοιχείο της στήριξης των στόχων της Ευρώπης 2020. κυρία Μαρία Αρενά μας επεσήμανε τα κριτήρια που θα πρέπει να είναι πανευρωπαϊκά. Αυτό είναι επίσης σημαντικό, το λέω και εγώ. Εγώ πάντως είμαι υπέρ της κινητικότητας. Γνωρίζω μάλιστα ότι ορισμένοι ευρωβουλευτές δυσαρεστούνται και δεν τους αρέσω ακριβώς για το λόγο αυτό. Νομίζω όμως ότι είναι σημαντικό διότι η κινητικότητα με υπευθυνότητα μπορεί να αποδειχτεί πάρα πολύ χρήσιμη. Μιλήσατε και για κοινωνική καινοτομία και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο διότι συχνά αντιμετωπίζω καταστάσεις όπου ορισμένοι δεν μπορούν να κατανοήσουν τι είναι κοινωνική καινοτομία. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. Ο συνάδελφός μου Τόμας Μαν, βεβαίω, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας κύριε Μαν, ότι για να μπορέσει να εφαρμοστεί το σχέδιο και να αποδώσει αποτελέσματα χρειάζεται ασφάλεια, εγγύηση των επενδύσεων γιατί έχουμε σήμερα δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία είναι παγωμένα, δεν τα χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις. Και γιατί, διότι δεν αισθάνονται ασφαλείς. Άρα πρέπει να είναι εγγυημένη η ασφάλεια των ε, επενδύσεων. να μπορούμε επίσης να αντιδράσουμε σε σφάλματα που μπορούν να γίνουν, να αλλάξουμε ό,τι χρειάζεται να αλλάξει και ούτω καθεξής. Δεν είναι πάντα αναγκαίο να περάσει μια πενταετία για να δούμε πώς λειτουργεί ένα εργαλείο που διαθέτουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν και αναμένω καρποφόρα συνεργασία. Ε, ευχαριστώ κυρία Γιασλοβιέτσκα. Το προσωρινό λοιπόν χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής για τις στρατηγικές επενδύσεις. Εξέταση του σχεδίου γνωμοδοτήσεως στις 5 Τρίτου. Κατάθεση τροπολογιών 6 Τρίτου. Έγκριση 1η Απριλίου 2015. Το τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξή μας, πριν από τη διακοπή του μεσημεριανού γεύματος, είναι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών μετά το 2015. Το λόγο θα δώσω αμέσως στην εισηγήτρια κυρία Κοσλόφσκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Η στρατηγική για την ισότητα ανδρών και γυναικών μετά το 2015 είναι κάτι το οποίο κοιτάει η Επιτροπή Γυναικών με μια σοσιαλίστρια για εισηγήτρια και βεβαίως η στρατηγική αναπτύσσεται με τακτικές συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους, ε, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί έχουμε πολλές διαβουλεύσεις, κάτι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ συχνό. Αλλά βεβαίως ε, μας βοηθάει όταν μιλάμε για να καταλήξουμε σε ένα έγγραφο το οποίο θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας. Μιλάμε λοιπόν για το τι γίνεται στην αγορά εργασίας, ε, το μέχρι που μπορούν να εξελιχθούν οι γυναίκες, ε, φτώχεια, βία κατά των γυναικών, ε, παρουσία τους στην αγορά εργασίας κτλ. Θα μιλήσουμε για τη δημογραφική κρίση και τη σχέση μεταξύ αγοράς εργασίας και την δυνατότητα να έχει κανείς τη δική της επιχείρηση αλλά και για τα ίσα δικαιώματα, η πτυχή δηλαδή εκείνη που αφορά την δυνατότητα να έχει κανείς μια επιχείρηση. Θέλουμε λοιπόν να προτείνουμε τα εξής πρώτον, δημογραφικό, σύμφωνα με πολλούς η δημογραφική κρίση σημαίνει πως οι δομές ε, της κοινωνίας και της οικογένειας αλλάζουν επίσης υπάρχουν επιπτώσεις στην αγορά εργασίας υπάρχουν λιγότεροι εργαζόμενοι στη χώρα μου στην Πολωνία υπολογίζεται πως μέχρι το 2035 εργαζόμενοι, ο αριθμός των εργαζομένων θα μειωθεί κατά 4 εκατομμύρια. Παρόμοιες αξιολογήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση λένε πως θα χάσουμε 24 εκατομμύρια εργαζόμενους μέχρι το 2040. Οπότε, για να αντιμετωπίσουμε την ε, πρόκληση αυτή θα πρέπει να μπουν στην αγορά εργασίας ε, οι γυναίκες. Υπάρχει μια διαφορά στη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας κατά 10-12% ίσως και παραπάνω. Και βεβαίως εκεί όπου αυξάνεται η συμμετοχή των γυναικών υπάρχουν περισσότεροι εργαζόμενοι. Ε, είναι λοιπόν σαφές πως ε, έτσι δεν θα έχουμε έλλειψη εργαζομένων. Οπότε είναι σαφές πως ε, η ισότητα των φύλων είναι βασική προϋπόθεση για να επιτύχουμε τον στόχο μας, δηλαδή ένα επίπεδο απασχόλησης της 100. Αν πετύχουμε αυτό το στόχο και δεν λέω ότι θα είναι εύκολο, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τις ε, ομάδες αυτές και θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος ε, στη συμμετοχή των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Το σημείο 3. Τονίζω πως η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα στην Ένωση εξαρτάται από το να καλυφθεί το χάσμα στην εκπαίδευση των γυναικών και στη συμμετοχή τους ε, στην αγορά εργασίας. Αν δεν σπάσει λοιπόν ε, αυτή η διαφορά, δηλαδή το πόσες είναι εκπαιδευμένες γυναίκες και το πόσες γυναίκες είναι σε διευθυντικές θέσεις ε, θα χάνουμε ταλέντο, θα πηγαίνει ανεκμετάλλευτο και θα σπαταλάμε και τα λεφτά τα οποία εξοδεύονται για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των γυναικών. Και αυτό λοιπόν πρέπει να συμπεριληφθεί στην έκθεση. Στο σημείο 4 τώρα μιλάω για τις αιτίες της ε, χαμηλής ε, συμμετοχής ε, των γυναικών. Δηλαδή βλέπουμε ότι σηκώνουν δυσανάλογο βάρος των οικογενειακών βαρών. Είναι ασύμετρη η κατάσταση στον οικοκυριό. Πρέπει λοιπόν να δούμε το τι γίνεται στις υπηρεσίες που καλύπτουν ε, αυτά τα ζητήματα, δηλαδή η φροντίδα των ηλικιωμένων, ε, των ασθενών, ε, βεβαίω παιδικούς σταθμούς και τέτοια πράγματα για να μπορούν οι γυναίκες να έχουν και προσωπική και οικογενειακή ζωή. και μία ισορροπία μεταξύ των δύο. Στο σημείο 5 μιλάω για την... τον εκθυλισμό της φτώχειας, την εκθύλυνση. Δηλαδή ότι οι γυναίκες είναι φτωχές και έχουν λιγότερα ένσημα και χαμηλότερους μισθούς και άρα χαμηλότερες συντάξεις τελικά. Ειδικά οι ηλικιωμένες γυναίκες λοιπόν είναι πιο φτωχές. Όταν ζουν σε ένα νοικοκυριό του ενός ατόμου και κάτι πρέπει να γίνει. Γιατί μιλάμε για εξάλληψη της στόχης μέχρι το 2020 και με όλες αυτές τις στρατηγικές πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, ακριβώς ε, τη γυναική φτώχεια, αλλιώς δεν έχουν κανένα νόημα. Επίσης για την άνηση μεταχείριση ανδρών και γυναικών θα καταπολεμήσουμε έτσι το πρόβλημα αυτό της φτώχειας. Στο σημείο 6 μιλάμε για την αναγκαιότητα μεγαλύτερης διαφάνειας ε, όταν ε, προσλαμβάνονται γυναίκες ε, σε διευθυντικές θέσεις. Εδώ πέρα υπάρχουν κάποια θετικά βήματα, αλλά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ακριβώς την ε, θέση των γυναικών και με διαφανείς ε, διαδικασίες να τις προωθήσουμε στις ε, διευθυντικές θέσεις. Στο σημείο 7. Στο σημείο 7 μιλάω για ένα πολύ συχνό φαινόμενο. Είναι η ανεπίσημη εργασία. Ήθελα λοιπόν να δημιουργηθεί ένα σύστημα κινήτρων για τους εργοδότες για να περάσουν οι γυναίκες από την ανεπίσημη στην επίσημη εργασία. Αυτά τα ολίγα, γιατί πρέπει να είναι σύντομη η γνωμοδότησή μου. Θα παρουσιάσω κάποιες τροπολογίες θα μιλήσω για ισότητα και ΑΕΠ, το χάσμα σε μισθούς και συντάξεις, για την εκπαίδευση και για το πώς θα καταπολεμήσουμε την άνηση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, ακριβώς για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα στην αγορά εργασίας. Και στο μέλλον θα καταθέσουμε και τροπολογίες ε, για ποσοστώσεις γυναικών σε διευθυντικές θέσεις. Και βεβαίως για τις δημόσιες προμήθειες. Ε, όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες, ξέρουμε πώς μπορεί να είναι αποτελεσματικές για να προωθήσουμε την κοινωνική πολιτική και την πολιτική κοινωνικής ένταξης. Μπορούμε λοιπόν να βάλουμε κάποιες κοινωνικές ρήτρε που με τη σειρά τους θα μας επιτρέψουν να δημιουργήσουμε περαιτέρω απαιτήσει για τις εταιρείες που θα πρέπει να εκπληρώνονται για να μπορεί η εταιρεία να υποβάλει προσφορές για δημοσιάργα. Στην Πολωνία έχουμε τέτοιες ρήτρε. Π.χ. κάποια έργα δίνονται μόνο σε, λεγόμενες, σε λεγόμενους κοινωνικούς συνεταιρισμούς ε, που απασχολούν δηλαδή κόσμο με αναπηρίες. Ή παραδείγματο χάρη ναι, μπορούμε να έχουμε μια απέτηση μια συγκεκριμένη εταιρεία να απασχολεί τουλάχιστον έναν ανάπηρο για να αναλάβει κάποια έργα. Ε, αυτές οι ρήτρε βεβαίως μπορούν να ισχύσουν μόνο εάν στα κρατη υπάρχουν σχετικοί κανόνες. και δεν υπάρχουν σε όλες τις χώρες ε, ε, κανόνες για ποσοστώσεις γυναικών σε διευθυντικές θέσεις. Όπου λοιπόν σπαταλάμε το χρήμα του φορολογουμένου μπορούμε να προωθήσουμε εταιρείες ε, οι οποίες ε, πληρώνουν όλες τις απαιτήσεις για ίση μεταχείριση ή να μπλοκάρουμε κάποιες εταιρείες από τη συμμετοχή στις δημόσιες προμήθειες αν παραβιάζουν τους σχετικούς κανονισμούς. Ε, αυτά είναι μόνο συστάσεις. Γιατί το θέμα είναι στα χέρια των κρατών μελών. Αλλά πρέπει παρόλα αυτά να πούμε τι σημαντικό εργαλείο μπορεί να είναι για να προωθηθεί ακριβώς μια τέτοια πολιτική. Αυτά από εμένα. Τώρα είμαι στη διάθεση των συναδέλφων για ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συναρπαστική ανασκόπηση. Ο λόγος στη Μαρία Ρενά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε για την ε, δουλειά που κάνατε συνάδελφε. Είναι μια πολύ καλή βάση εργασίας για αυτή τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης. Εξίσου σημαντικό είναι και αυτό το θέμα να απασχολήσει την Επιτροπή μας, διότι υπάρχει σοβαρή διακριτική μεταχείριση στην Ευρώπη κατά των γυναικών αυτή τη στιγμή και αφορούν οι μορφές αυτές διακριτικής μεταχείρισης ε, την ε, εργασία το θέμα της βίας που θα καλυφθεί στην έκθεση Νόιχλ είναι άλλο βέβαια, αλλά το βασικότερο που μας απασχολεί εδώ σήμερα είναι το τι συμβαίνει στον εργασιακό χώρο. Γι' αυτό έχω επιτρέψει τον εαυτό μου να υποβάλει κάποιες τροπολογίες, θα αναφέρω μόνο μερικές σήμερα, για να βελτιώσω λίγο το κείμενο. Πρώτον, να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι η ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας και το ποσοστό που έχουμε στόχο στο Horizon 2020, αλλά και για την καταπολέμηση της κρίσης, είναι ένας στόχος κοινωνικής δικαιοσύνης πάνω απ' όλα. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν υπήρχε κρίση, ακόμα και αν πήγαιναν τέλεια σε έναν ιδανικό κόσμο, θα υπήρχε ε, πρόβλημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Πρέπει λοιπόν να το θυμίσουμε. Δεύτερον, το περίφημα ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών 50% έως το 2020 και, το στόχο, για το στόχο μείωση τη φτώχεια. Ξέρουμε ότι οι γυναίκες ε, στην εργασία, εάν μιλάμε για εργασία ποιότητα, αυτό το δούμε στο σημείο 3, οι, γυναίκες πρέπει να βρεθούν σε θέση λιγότερη εξάρτηση και λιγότερη φτώχεια. 20% των πολιτών τη Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι φτωχοί. Τρίτο σημείο, και το είπα, είναι η εργασία ποιότητα. Ε, Δυστυχώ, αν δει τα στατιστικά στοιχεία, οι γυναίκε πλήττονται περισσότερο από την επισφαλή εργασία, από αυτό το σύστημα, από την αδήλωτη, την ανεπίσημη εργασία. Είναι λοιπόν σημαντικό να εργαστούμε για την ποιότητα της εργασίας και έτσι περνάω στο τέσσερα. Ποιότητα της εργασίας για τις γυναίκες σε μια περίοδο συγκεκριμένη της ζωής τους το, την άδεια μητρότητας. Εδώ πρέπει να υπάρξει εξυγχρονισμένη νομοθεσία στην Ευρώπη που να ισχύει παντού για την άδεια μητρότητας. Οι γυναίκες αυτές πρέπει να προστατεύονται τη στιγμή που κυοφορούν και τη στιγμή που μόλις έχουν ε, περάσει από το δοκετό ε, και δεν είναι στην αγορά εργασία. Πρέπει λοιπόν και από δημογραφική άποψη να δούμε το θέμα τη άδεια μητρότητα, διότι είτε θα αποκτήσουμε γυναίκε που δεν θα θέλουν πια να κάνουν παιδιά και ήδη τα ποσοστά γεννήσεων σε πολλέ χώρε ε, έχουν πάρει την κατιούσα, είτε γυναίκε που δεν θα πηγαίνουν να δουλέψουν, διότι δεν θα έχουν καμία ασφάλεια. Πρέπει ε, πάση θυσία να υπάρξει μια εκφρονισμένη νομοθεσία για το θέμα. Και επίση μια νομοθεσία που να επιτρέπει να συνδυαστεί καλύτερα επαγγελματικό με τον επαγγελματικό βίο και να επιμεριστεί καλύτερα ο φόρτο εργασία μεταξύ ε, των ανδρών και των γυναικών στο ρόλο του πατέρα και τη μητέρα. Είναι σημαντικό και αυτό από την προοπτική τη απασχόληση. Τελευταία μέρημνα, ε, όχι τελευταία, μία από τι σημαντικέ ενώ, είναι η εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Ξέρετε ότι σήμερα γίνονται ήδη συζητήσει, μπορούμε να έχουμε καλές προθέσεις λέγοντας ότι θέλουμε περισσότερες γυναίκες ε, αλλά όταν μιλάμε για δεσμευτικούς νόμους ακούω κάποιοι να έχουν επιφυλάξεις και να μην θέλουν να πιέσουν τι επιχειρήσει να έχουν περισσότερε γυναίκε στα διοικητικά συμβούλια. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα λόγο να μην υπάρχουν περισσότερε γυναίκε. Είναι πιο ε, ψηλά τα ποσότητα των γυναικών σήμερα κατά μέσο όρο. Έχουν περισσότερε σπουδέ και πτυχία από ότι άντρε. Εκπροσωπούνται στι γυναίκε, στι επιχειρήσει, συγγνώμη. Το να ε, συμμετέχει μια γυναίκα σε διοικητικό συμβούλιο δεν κοστίζει περισσότερο από ότι να συμμετέχει ένα άντρα. Δεν υπάρχει πρόβλημα κόστου ούτε δεξιοτήτων. Το μόνο πρόβλημα είναι ο συντηρητισμό των ανδρών που σκέφτονται ότι μια γυναίκα θα αντικαταστήσει έναν άντρα. Αυτό πρέπει να το πολεμήσουμε. Οι γυναίκες να εκπροσωπούνται με ποσοστώσεις στα δικαιωτικά συμφόλια για να αλλάξουν λίγο, να αναταραχθούν και να μετακινηθούν οι καθεστικέ συμπεριφορές. Ε, Ευχαριστούμε. Η Τάνια Γκονσάλες Πένιας είναι εδώ. Αφού διάβασα τις ε, προτάσεις ε, της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών, πρέπει να πω ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά στοιχεία για να πετύχουμε περισσότερη ισότητα. Ε, είναι σημαντικό να τονίσουμε τη σημασία της σωστής κατανομής του φορτοεργασίας. μια διεκδίκηση που ήδη γίνεται στην αγορά εργασίας για τα ωράρια και τη φροντίδα των παιδιών. Επίσης, τα, οι συμβάσεις μερικής εργασίας, προσωρινής εργασίας για τις γυναίκες πρέπει να επανεξεταστούν για να υπάρχει ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Πρέπει να δούμε επίσης και τις δομές και υπηρεσίες ε, αρρωγής και στήριξης. Αλλά να υπάρχει και εκπαίδευση, νηπιακή εκπαίδευση από πολύ μικρή ηλικία με ταυτόχρονα υπηρεσίες για ηλικιωμένους που να είναι δημόσιες διαχείρισης. Επίσης, οι γυναίκες πολλές φορές ασχολούνται με την περίθαλψη άλλων προσώπων του περιγύρου τους και με πολύ κακές αμοιβέ και Ενώ πολλέ φορέ οι γυναίκε κάνουν την ίδια δουλειά με έναν άντρα, παίρνουν λιγότερε αμοιβέ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να απολωμήσουμε ε, με τρόπο ε, δραστικό την ε, μισθολογική μορφή διακρίσεων. Όταν μιλάμε για υπεύθυνη πατρότητα και αύξηση των αδειών, εδώ νομίζω σημαντικό είναι η άδεια πατρότητας να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα και αυτή της μητρότητας ώστε να είναι ίσες και να εξασφαλίσουμε άδειε μητρότητας και πατρότητας ε, ώστε να μπορούν να ε, μεγαλώνουν οι οικογένειες. Αυτό μου φαίνεται ένα σημείο κλειδί στο έγγραφο και, στο έγγραφο και να μην ξεχνάμε το θέμα της φτώχειας. Είναι σημαντικό να θυμάμαστε ότι οι γυναίκες έχουν περισσότερα ποσοστά φτώχειας και ότι υπάρχουν ε, σοβαροί λόγοι που εξηγούν γιατί αυτό συμβαίνει. Όμως σημαντικό είναι ότι οι γυναίκες πολλές φορές δουλεύουν εκτός ωραρίων με κακές αμοιβέ και με λιγότερα συνταξιδοτικά δικαιώματα. Ακόμη λοιπόν και από την προοπτική των συντάξεων που δεν έχουν σωρευτική διάσταση, πρέπει να βρεθεί μια λύση για να αντιμετωπίσουμε την φτώχεια και ε, για τις γυναίκες και την παρουσία τους στα διοικητικά συμβούλια και στη δικασία λήψη αποφάσεων. Αυτό δεν πρέπει να ισχύει μόνο για τις επιχειρήσεις αλλά και για, τα, για τους δημόσιους φορείς και γενικώ σε οποιοδήποτε επαγγελματικό κλάδο. Οι γυναίκες πρέπει να είναι σε τέτοιες θέσεις που να μπορούν να λάβουν αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα ε, και στο πολιτικό. Οι δημοσίες υπηρεσίες έχουν σοβαρές επιπτώσεις ε, στη ζωή των γυναικών ανάλογα με το πώς προσφέρονται. Δηλαδή, Πριν τις περικοπές ε, σε ορισμένε χώρες της Ευρώπης υπήρχε μεγάλη παρουσία των γυναικών στις δημόσιες υπηρεσίες. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν και πάλι ισορροπία στην αγορά. Πρέπει να σταματήσουν οι περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες διότι πορεία προς τη φτώχεια και η ανισότητα θα συνεχιστούν. Πιστεύω ότι οι προτάσεις για ορισμένα από τα στοιχεία του εγγράφου ε, από την Επιτροπή Ισότητας και γυναικών ε, είναι τροπολογίες που θα πρέπει να διατηρηθούν. Ε, απλώς πρέπει να διευκρινίσουμε ποια είναι τα γενεσιουργά αίτια της ανισότητας ανδρών και γυναικών. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια για την σύνταξη της έκθεσης αυτής. Γνωρίζουμε ότι η ισότητα των φύλων δεν θα ωφελήσουμε τι γυναίκε εάν βελτιωθεί η κοινωνική και η οικονομική ευημερία, αλλά όλη την κοινωνία. Η ισότητα των φίλων από τι αρχέ τη τις της Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν μια από τι θεμελιώδει μα αρχέ και αξίε. Ήδη πριν από 50 χρόνια η αρχή τη ίση αμοιβή ήταν κάτι που εγγράφει στι συνθήκε. Αυτό είναι σκανδαλώδε να μην έχουμε ακόμα σήμερα στην πραγματικότητα ίσε αμοιβέ μεταξύ άντρων και γυναικών, Ίσες, ε, παρόμοιε προποθέσει για άντρε και γυναίκε στην αγορά εργασία. Ω πρώτα τη στρατηγική ισότητα των φύλων, βλέπουμε πολλέ κρίσιμε πτυχέ για την ζωή των γυναικών, για το χάσμα των αμοιβών, για την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών, για την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασία και τη σταδιοδρομία του, για την ίση εκπροσώπηση στη διαδικασία λήψη αποφάσεων και για την άρση των διακριτικών μεταχειρήσεων και των μορφών διακριτική συμπεριφορά σε σχέση με τα θέματα του φύλου. Όλα αυτά είναι κέρια σημασία. Να ε, πιστήσω την προσοχή σα σε ένα-δυο σημεία που ε, έδωσαν και το πνεύμα στι τροπολογίε που υποβάλαμε. Πρώτα απ' όλα, ε, ο εκτεθλισμό τη φτώχεια. Εδώ πιστεύουμε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα πολλών συνδυασμένων παραγόντων, όπως του χάσματος των αμοιβών που κάνει πιο δραματικό και το συνταξιωτικό χάσμα ή της περιπτώσεις ε, περίθαλψης που πολλές φορές αναβαλάμαν οι γυναίκες. Το κοινωνικό σύστημα ή τα φορολογικά συστήματα. Εγώ έρχομαι από μια χώρα που το φορολογικό σύστημα είναι λόγος να υπάρχει μεγαλύτερη ανισότητα ανδρών και γυναικών. Η καταπολέμηση της φτώχειας ε, 20 εκατομμύρια έως το 2020 είναι κάτι που μπορεί να ε, επιληθεί μόνο με την ευθυγράμμιση των φύλων σε όλες τις πολιτικές και με την στοχοθέτηση της γυναικείας φτώχειας. Εάν οι γυναίκες δεν είναι πρώτες σε αυτόν τον αγώνα, δεν θα φτάσουμε τους στόχους μας. Αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τα μέτρα λιτότητας στην Νότια Ευρώπη είναι ότι υπήρξε μια αντίστροφη εξέλιξη. Οι γυναίκες έχουν πληγεί πέρμετρα από τα μέτρα αυτά. Εάν δει κανείς την πραγματικότητα των γυναικών καταλαβαίνει ότι τα μέτρα λιτότητας είχαν αρνητικό αντίκτυπο και ότι χρειαζόμαστε στο μέλλον να αγωνιστούμε για να μην γίνει ακόμα χειρότερη κατάσταση. Η τελευταία μου παρατήρηση και επειδή έχουμε υποβάλει τροπολογίες για το θέμα αυτό αφορά την σεξουαλική παρενόχληση ε, στην εργασία αλλά και την ομοφοβία καθώς και την ε, φοβία των διαφυλικών στον χώρο εργασίας. Η στρατηγική για την ισότητα των φύλων πρέπει να λάβει υπόψη και την ταυτότητα των φύλων και την ε, φοβία προς τους λαόδι υπόψη, γιατί είναι ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να καλύψουμε. Ευχαριστούμε Τιτσιάνα Μπεγκίν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την ε, εισηγήτρια για την έκθεσή της. Είναι σημεία όλα πολύ σημαντικά και τα συμμεριζόμαστε. Απλώς να δώσω έμφαση στο γεγονός ότι προφανώς το πρόγραμμα συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι ένα πρόβλημα σοβαρότατο. Για να το επιλύσουμε θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα γενεσιουργά αίτια. Νομίζω ότι ακόμα σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολύ συχνά ζητάτε από τις γυναίκες να διαλέξουν μεταξύ δουλειά και οικογένειας. Πάρα πολύ συχνά αυτό εμποδίζει την πρόσβασή του στην αγορά εργασίας και πολλές φορές δεν σκεφτόμαστε πώς να διευκολύνουμε την επανένταξή του στην αγορά εργασίας. Το λέω ως μητέρα, κόρη και ε, εργαζόμενοι σε μεγάλες επιχειρήσεις στην Ιταλία. Οι διακρίσεις ε, στην, στο χώρο εργασίας υπάρχουν ακόμη και πολλές φορές προτιμώνται υποψήφοι άντρες για τις θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν. Στις γυναίκες ε, τέθενται ερωτήσει όπως πώς θα συνεχίσουν να δουλεύουν μετά το γάμο, πώς το σκέφτονται και ενώ είναι νόμιμα όλα αυτά συνεχίζονται αμύωτα. Η συμπεριφορά προς τις γυναίκες, η συμπεριφορά που επικρατεί, όπως υπογράμμισαν και οι συνάδελφοι, δυστυχώς συχνά είναι στερείται αξιοπρέπειας για να μην φτάσουμε να μιλήσουμε για παρενόχληση, αλλά η διάκριση σε καθημερινό επίπεδο είναι σύνηθες φαινόμενο. Ε, και από τη μισθολογική πλευρά και από τη συνταξιδοτική. Με λύπη μου λέω πως η χώρα μου είναι από τις τελευταίες της υπηρεσίες προς τις οικογένειες, αλλά κανείς στην Ευρώπη δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν υπάρχει στη χώρα του το πρόβλημα αυτό. Υπάρχει μια πολύ ανδροκατούμενη νοοτροπία ακόμη στην Ευρώπη. Οι υπηρεσίες προς την οικογένεια λοιπόν ε, ε, είναι κάτι που αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου γυναίκε και συχνά χρειάζεται να απαρνηθούν την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Δεν επιστρέφουν καν στην ε, εργασία του μετά από μία εγκυμοσύνη ή δεν προχωρούν στη σταδιοδρομία για να ασχοληθούν με την ανατροφή των παιδιών του. Το λέω ω ε, από προσωπική πείρα, διότι όταν έχει κανείς παιδιά δεν κάνει θανάσιμα άλματα δεν αναλαμβάνει ρίσκα. Ε, βέβαια, το πρόβλημα δεν είναι μόνο νομοθετικό, είναι και πολιτιστικό χαρακτήρα, νοοτροπία. Αλλά πρέπει εδώ να έχουμε μια αποτελεσματική τοποθέτηση ω θεσμικά όργανα. Ε, είναι η περίοδος της αποτελεσματικής χρήσης των ε, πόρων. Ένα από, μια, ένας από τους σημαντικότερους πόρους που δεν έχουμε αξιοποιήσει ακόμα επαρκώς είναι οι γυναίκες. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρώπη και τα κάτι μέλη πρέπει να δράσουν για να σταματήσει αυτή η αρνητική πορεία. Ευχαριστώ. Thank you. Η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ, κυρία Σαρτή. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Έχουμε ένα θέμα που μας απασχολεί έντονα, βέβαια και μέσα στις συνθήκες που βρισκόμαστε. Θα ήθελα λοιπόν πρώτα να θέσω επιτάπητος τρία δεδομένα που είναι πολύ σημαντικά. Την επίπτωση της κρίσης στην ε, εργασία των γυναικών. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο η επίπτωση της κρίσης στην εργασία των γυναικών έδιωξε τις γυναίκες από την αγορά εργασίας που υποπληρώνονταν αβέβαιες εργασίες μερικού χρόνου, ακόμα χειρότερο όμως. Όχι μόνο η κρίση ανάγκασε τις γυναίκες να φύγουν από τις δουλειές, αλλά οι γυναίκες ενέτειναν την κίνηση αυτή εν ώψη και της δυσκολίας να εξασφαλίσουν την ισορροπία ανάμεσα στην οικογενειακή ζωή και στην επαγγελματική ζωή, εγκατέλειψαν λοιπόν την ε, αμοιβόμενη εργασία και πήγαν σε ε, εργασίες μη αμοιβόμενες. Και αυτό, αυτή η κίνηση έχει ενταθεί από την κρίση. Πρέπει να εμείνουμε σε αυτήν την διεύρυνση των ανισοτήτων ανδρών και γυναικών μέσα στη δουλειά που συνδέεται με την κρίση. Δεύτερο στοιχείο είναι αυτό της νοοτροπίας που οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε. Στη χώρα μου κάναμε μια δημοσκόπηση που περιείχε την εξής ερώτηση. Θεωρείτε ότι σε περιόδους κρίσεων οι άνδρες πρέπει να έχουν προτεραιότητα στην έβρεση εργασίας και χαίρομαι που με ακούνε και οι σοσιαλίστρες. Πρέπει λοιπόν να έχουν προτεραιότητα στην έβρεση εργασίας. 63% των ερωτηθέντων είπαν ναι. Να λοιπόν ένα πραγματικό πρόβλημα νοοτροπίας που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Σε αυτά τα 63% των ερωτηθέντων υπάρχουν και ερωτηθήσεις. Πρέπει να σπάσουμε αυτή τη γυάλινη οροφή, πρέπει δηλαδή να βρίσκουμε τις γυναίκες να σπάσουν τη γυάλινη οροφή. Και το τρίτο είναι η εκπαίδευση, κάτι είπατε σχετικά, που αποτελεί σημαντική επένδυση και δημόσια και ιδιωτική. Εκπαίδευση και από την πλευρά των κρατών και από την πλευρά των οικογενειών. Δεν υπάρχει βέβαια απόδοση της επένδυσης αυτής στον τομέα της εργασίας. Εγώ θα κάνω βεβαίως κάποιες σχετικές τροπολογίες. Μια πραγματική κινητοποίηση, διότι συμφωνούμε πολλά από όσα λέγονται, από όσα γράφονται μέσα στη γνωμοδότηση. Βλέπω όμως να λείπει ο αγώνας κατά των ανισοτήτων στις σταδιοδρομίες. Βεβαίως υπάρχουν ανισότητες αμοιβών. Αν όμως περιοριστούμε μόνο στην ανισότητα των αμοιβών ή των μισθών, ποτέ δεν θα φτάσουμε σε, σε αυτή την πραγματική απορρόφηση, αντιμετώπιση των ανισορροπιών. Διότι υπάρχουν ανισότητες στην σταδιοδρομική εξέλιξη που αναγκάζουν τις γυναίκες να παραμείνουν στη φτώχεια στην πραγματικότητα, διότι μια γυναίκα που φτάνει σε τη συνταξιωτική ηλικία λαμβάνει το 37% του ε, μισθού του άνδρα. Δεύτερο, που θα πρέπει να γίνει κάποια σχετική τροπολογία, είναι οι ανισότητες για τα κριτήρια πρόσληψης. Στην έκθεση που έκανα εγώ για την ε, επίπτωση της κρίσης ε, στην εργασία των γυναικών, διαπιστώνουμε ότι το πρώτο κριτήριο πρόσληψης για μια γυναίκα είναι η διαθεσιμότητα. Οι ικανότητες, δεξιότητες έρχονται σε δεύτερη θέση, ενώ πρώτο κριτήριο πρόσληψης για έναν άντρα είναι οι δεξιότητες. Η διαθεσιμότητα έρχεται δεύτερη. Έχουμε δηλαδή ακριβώς ένα σχήμα χιαστή. Τα κριτήρια πρόσληψης μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι ακριβώς αντίθετα. Άρα, νοοτροπίες, κριτήρια πρόσληψης, ανισότητες στη σταδιοδρομία αποτελούν θεμέλια που πρέπει να ανατινάξουμε για να μπορέσουμε να φτάσουμε να οικοδομήσουμε μια ισότητα μεταξύ άνδρων και γυναικών. Άκουσα την Μαρία Αρένα πριν να μιλεί για το πρόβλημα της μητρότητας και την επίπτωση στην σταδιοδρομία της γυναίκας. Λυπούμε όμως που δεν εναρμονίσαμε σε επίπεδο των 28 χωρών μελών στην προηγούμενη κοινοβουλευτική μας θητεία τις ε, άδειες μητρότητας, όπως λέω, και σε όλες τις ε, ε χώρες μέλη. Πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό, να μην προσπαθούμε να επιτύχουμε στόχους που δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν. Να συμφωνήσουμε όπως στην ουσία τα είχαμε καταφέρει να συμφωνήσουμε πάνω σε, μια ε, αμοιβόμενη άδεια μητρότητα στις τάξεις των 16-18 ε, ε, εβδομάδων. Γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν 56 εβδομάδες αλλά μη αμοιβόμενες. Πέραν λοιπόν όλων των κομμάτων, πέραν όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων, να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτή τη συμφωνία. Διότι αν δεν τα καταφέρουμε εδώ, τότε όλοι οι αγώνες μας, όλες οι μάχες μας είναι εισμάτιν. Σε ό,τι αφορά τις ποσοστώσεις, εγώ ήμουν αντίθετη και αγωνίστηκα κατά αυτόν εδώ και μια δεκαετία, το 2000, αρχές του 2000. Διότι θεωρώ ότι με τις ικανότητές τους, με τις δεξιότητές τους, οι γυναίκες μπορούν να τα καταφέρουν. Όμως τώρα μια δεκαετία μετά αντιλαμβάνομαι ότι οι ικανότητες όσες και τα προσόντα όσα και να έχουν οι γυναίκες δεν αρκούν. Και αν δεν βάλουμε ποσοστώσεις δεν πρόκειται ποτέ να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Για μένα λοιπόν είναι υποχρεωτική η διέλευση από αυτό. Ελπίζω δηλαδή κάποια στιγμή να μπορούμε να πούμε ότι κάναμε τόσο καλά τη δουλειά μας ώστε να μην έχουμε πλέον ανάγκη ποσοστώσεων. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η ε, κυρία Πρόεδρος. Ευχαριστώ, κυρία Σοϊντέροβα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε το λόγο. Και χαίρομαι που λαμβάνω το λόγο μετά την κυρία Σορτιέ. Θα ήθελα να προσθέσω και εγώ κάποια πράγματα που θεωρώ σημαντικά. Κατά την άποψή μου η θέση των γυναικών βασίζονται στο ότι οι γυναίκες είναι απολύτως απαραίτητες για κάθε οικογένεια και δεν μπορεί να τις αντικαταστήσει κανείς σε αυτό το ρόλο. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως έχουν ένα εμπόδιο όταν θέλουν να επανέλθουν στη δουλειά, κάτι το οποίο ανέφεραν ήδη οι συνάδελφοι. Αυτό δεν είναι η εντύπωσή μας, ε, έτσι είναι η πραγματικότητα και το αποδεικνύει και μια έρευνα που έγινε το 2011-12, ΠΕΑΚ λέγεται, μία μελέτη του ΟΣΑ που βασίζεται στην αγορά εργασίας η οποία έδειξε πως οι γυναίκες ε, μετά την άδεια μητρότητας ε, έχουν ε, νέες ικανότητες αλλά παραδείγματος χάρη μένουν πίσω σε σχέση με τους άντρες ε, όταν επιστρέφουν από την ε, άδεια μετρότητα. όταν μιλάμε για ε, δεξιότητες στον τομέα της πληροφορικής. Δηλαδή πανέρχονται στην αγορά εργασίας γύρω στα 30, η σημαντικότερη κατηγορία Η συνάδελφος ανέφερε επίσης πως στην έρευνα ήταν σαφές πως ο κόσμος προτιμάει άνδρες σε αυτές τις θέσεις. Και φαίνεται και φυσικό οι εργοδότες να προσλαμβάνουν άνδρες γιατί θεωρούν πως οι άνδρες είναι πιο διαθέσιμοι και ότι θα έχουν ε, μεγαλύτερη σταδιοδρομία και άρα ταιριάζουν καλύτερα σε αυτές τις θέσεις. Πρέπει να εστιάσουμε λοιπόν στην περίοδο στην οποία οι άνδρες επανέρχονται οι γυναίκες με συγχωρείτε επανέρχονται στη δουλειά μετά την άδεια μητρότητας. Πρέπει λοιπόν να τις στηρίξουμε για να επανέλθουν ή να τις στηρίξουμε για να ξεκινήσουν την δική τους εταιρεία. Αυτό είναι το βασικό, να μην γίνονται διακρίσεις Επίσης, ε, κατά την άποψή μου, πρέπει να ε, υπάρχει περισσότερη στήριξη για τηλεεργασία και τα λοιπά. Περισσότερη στήριξη λοιπόν για τις γυναίκες που επανέρχονται στην αγορά εργασίας μετά από την άδεια μητρότητας. Επίσης είναι άδεια μητρότητας. Ε, δεν είναι άδεια όμως, δεν κάθεται. Δηλαδή η γυναίκα δουλεύει συνέχεια με τα παιδιά της και πρέπει να το σεβαστεί αυτό η κοινωνία. Σας ευχαριστώ. Η Κομισιόν είναι ακόμα εδώ. Ωραία. Θέλετε να πείτε λίγα λόγια. Έχετε τον λόγο. Κυρία Πετάκ. Γεια σας. Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να τονίσω πρώτα απ' όλα πως αυτό το αυτά τα οποία λέτε αναφέρονται ήδη στην τρέχουσα στρατηγική για την ισότητα των φύλων. Κάποια άλλα τα γνωρίζουμε αρκετά καλά, γνωρίζουμε πως πρέπει να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο στο μέλλον και γνωρίζετε πως αναμένουμε τη νέα στρατηγική τον Απρίλιο και αναμένουμε ιδέες, συλλέγουμε ιδέες. Θα μεταφέρω αυτά τα οποία είπατε στους συναδέλφους μου και βέβαια συμφωνούμε πλήρως με όλες τις παρατηρήσεις σας. Νομίζω πως οι περισσότερες ιδέες σας που αφορούν την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και η πιο σημαντική προτεραιότητα είναι αυτή και θα συνεχίσουμε έτσι και στο μέλλον. Καλώς ορίζω λοιπόν τα σχόλιά σας, συμφωνούμε πλήρως και όπως είπα θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα αυτά τα ζητήματα που δεν ε, τα είδαμε ίσως τόσο πολύ στην τωρινή στρατηγική όπως τη φτώχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό. Σας ευχαριστώ. Κυρία Κοσλόφσκα, έχετε λίγα λόγια και εσείς να πείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα και εγώ να πω το εξής. Είναι σαφές πως ε, η άνηση μεταχείριση και τα στερεότυπα δεν ε, κάνουν μόνο τις γυναίκες πιο φτωχές, αλλά εμποδίζουν και την οικονομική ανάπτυξη. Οι περισσότερες παρατηρήσεις που έγιναν αφορούσαν ζητήματα που είναι ήδη στην ε, έκθεση, οπότε πρέπει να τα τονίσουμε ίσως ξανά. Αλλά προέκυψαν νέα δεδομένα στην συζήτηση που θα περιληφθούν νομίζω στην γνωμοδότηση π.χ. ανεπίσημη εργασία από τις γυναίκες ε, πρέπει να δώσουμε περισσότερο βάρος σε αυτό. Βία επίσης παρενόχληση στη δουλειά, σεξουαλική παρενόχληση όπως επίσης και η απέτηση εναρμόνισης ε, των αδειών μητρότητας και πατρότητας. Πρέπει να προωθήσουμε τα δικαιώματα των ε, πατεράδων ε, και των μητέρων οπωσδήποτε. Οπότε εγώ δεν έχω πρόβλημα με τις άδειε ε, πατρότητας. Όσον αφορά τώρα την άνηση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας και τις διαφορετικές ε, αντιλήψεις που υπάρχουν, αυτά τα πράγματα είναι γνωστά, π.χ. στην ε, Πολωνία ε, υπήρχε μια γνωμοδότηση από την Παγκόσμια Τράπεζα και είχε γίνει μια έρευνα εκεί πέρα για την ιεραρχία και τις θέσεις που καταλαμβάνουν άνδρες και γυναίκες. Και οι άνδρες με παιδιά ε, θεωρούνται οι πιο αξιόπιστοι μετά οι ε, άνδρες ε, χωρίς παιδιά οι οποίοι ε, θεωρούνται πιο διαθέσιμοι. Οι γυναίκες παιδιά ήταν στον πάτο της λίστας γιατί θεωρούσαν πως ήταν υψηλού κινδύνου. Οπότε το να έχει παιδιά ο άντρας και η γυναίκα ε, το βλέπουν διαφορετικά οι εργοδότες. Γιατί τις γυναίκες τις συνδέουμε με την ανατροφή των παιδιών Κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα λείπουν πιο συχνά από τη δουλειά και αυτό σημαίνει πως οι εργοδότες θεωρούν ε, πως οι άνδρες και οι γυναίκες είναι διαθέσιμοι σε διαφορετικό βαθμό. Πρέπει να τα καταπολεμήσουμε αυτά τα στερεότυπα, αλλά και να βοηθήσουμε άνδρες ε, και γυναίκες να συνδυάζουν ε, οικογενειακή και επαγγελματική ζωή. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, θα υπάρχουν σοβαρές συνέπειες. Ε, εκτός, τι να πω, εάν ε, δεν, ε, εκτός να καταργήσουμε τη μητρότητα και τα παιδιά. Δεν το βλέπω πιθανό. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ.